Uh, um, Καλημέρα σας. Να σας ε, καλωσορίσω στην σημερινή συνεδρίαση. Ο λόγος για τη μεγάλη αίθουσα είναι η χθεσινή ακρόαση. Οπότε κάπως σήμερα κόντυνα τη λαλό μου, αλλά τι να κάνουμε. Μια ακόμη δύσκολη δουλειά μας περιμένει σήμερα και σημαντικές ψηφοφορίες και 9.30. Θα συζητήσουμε όμως πρώτα απ' όλα μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση. Όσοι ήθιστε, μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου η συνεδριασή μας. Ελπίζω να υπάρχουν πολύ ενδιαφερόμενοι για τις κλινικές δομικές. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι υπάρχει και η μηνία μας εφημερίδα. Τη βλέπετε. Μπορείτε να μας στείλετε ένα email, να γίνετε συνδρομητές και να μέσω email. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά στοιχεία σε αυτό το newsletter και πολλά έγγραφα σχετικά με το έργο μας. Σε ό,τι αφορά την πρόταση κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές, ο κύριος Ποσόη μας υπέβαλε τις τροπολογίες του και τώρα έχουμε, εφόσον εξετάσει την επίσημη πρόταση, εξετάζουμε και τις τροπολογίες των σκιωδών, τους οποίους καλημερίζω. Um, uh, uh, Και λοιποί έρχονται. Κυρία Μακλάρκιν, ούτε αυτή είναι εδώ. Ο Στέφανο Σόρο από την Κομισιόν, πολύ τακτικός μα επισκέπτης, να τον καλημερίσουμε και αυτόν. Θα του δώσουμε την ευκαιρία να πει και αυτό λίγα λόγια μετά. Αυτή η γνωμοδότηση θα περάσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι επικεφαλής, η αρμόδια δηλαδή Επιτροπή, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι σημαντικό να έχουμε κι λόγο για τη δημιουργία ενό πραγματικά αποτελεσματικού πλαισίου για τα φάρμακα των ασθενών. Πρώτα απ' όλα ο για το λόγο και μετά πάνω σκιώδε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Θα πω λίγα λόγια για τι δικέ μου τροπολογίε. Τι τροπολογίε των εισηγητών ευχαριστώ όσου υπέβαλαν τροπολογίε αυτόν τον χρονισμό ε, για τη συμβολή του στην όλη προσπάθεια. Σε τόση γνώμη Ε, λίγο πριν αρχίσουν οι ψηφοφορίε, 9 και 25 πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να προλάβω την πτήση μου για μια διάσκεψη στο Βουκουρέστι. Θα είμαι όμω ε, σύντομο και νομίζω ότι και οι ενδιαφερόμενοι σκιώδεις ε, έχουν να πούν πολλά ακόμη και θα έχουμε πιο πολλές συζητήσεις με την τελική ψηφόρια. Εν είδη γενικού σχολείου θα πω ευθύς εξ αρχής ότι ο στόχος μου είναι η διαδικασία να παραμείνει όσο γίνεται πιο απλή, ώστε να είναι και ταχύτερη. Κατανοώ ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ περιττικά για κάποια κράτη-μέλη κάποιοι μπορούν να τα βρουν και αδύνατο να τα επιτύχουν. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η ταχύτητα τη αδειοδότηση είναι στοιχείο κλειδί, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο διαλεστική για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών και να γίνει πιο στην κλινική έρευνα εν γέννη ο κανονισμός τώρα βασίζεται στην αρχή της σιωπηρής ε, συμφωνίας. Πολύ σημαντική διασφάλιση ώστε τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα. Οι εμπειρίες σχετικές από τις οδηγίες μας δείχνουν για ποιο λόγο είναι αυτό σημαντικό. Οπότε, εγώ δεν θέλω τροπολογίες που να θίγουν αυτή την αρχή. Στηρίζω όμως τη διευκρίνηση. Δηλαδή, αν κάποιο κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει αντίθετη γνώμη πριν την προθεσμία, θεωρείται ότι εγκρίνει την πρόταση του κανονισμού. Τώρα για τις επιτροπές διοντολογίας Ακόμα και αν δεν φέρουν αυτήν την ονομασία, θα υπάρχουν. Και οι πιο πολλοί σκιώδεις έχουν παρόμοια ανησυχία με μένα. Το θέμα λοιπόν είναι πού θα μπει αυτή η αφορά στις επιτροπές δεοντολογίας, ώστε να μην υπάρχουν επαναλήψεις και να υπάρχει ακολουθία στο κείμενο. Η τροπολογία που λέει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να διαφωνήσει για διδολογικά ζητήματα α, με το κράτος μέλος που κάνει την ενημέρωση και αναφορά. Αυτό πιστεύω είναι πολύ γενικό. Άρθρο 86, το οποίο αναφέρεται ήδη στην χρήση κάποιων κατηγοριών κιτάρων βάσει εθνικής νομοθεσίας, είναι επαρκής κλίδα ασφαλείας ε, και σε ό,τι αφορά τώρα κάτι άλλο για την ενημερωμένη συνένωση. Πιστεύω ότι υπάρχουν τα κατάλληλα εχέγγυα. Όμως, θα πρέπει να υπάρχει και περισσότερη ευελιξία ώστε να λάβουμε υπόψη το πώς πρακτικά γίνονται οι κλινικές δοκιμές και πώς άτομα ε, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ε, σε κάθε περιπτώση, ο κύριο Ζουβάν που είναι ειδικό σε αυτόν τον τομέα, μου έκανε πολύ ενδιαφέρουσε τροπολογίε. Κάποιε τροπολογίε πάντω χρήζουν πολύ προσοχή προσοχής ε, σε ό,τι αφορά την ενημερωμένη συνένεση. Η διαφάνεια σε πολλά σημεία του κειμένου είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρή υπόψη πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πού είναι απαραίτητη η διαφάνεια και πού δημιουργεί απλά εμπόδια. Για παράδειγμα, για την απόσταση μιας άδεια. Ε, η προτέρα διαβούλευση δεν έχει κάποιο νόημα. Ή όταν μια δοκιμή ολοκληρώνεται πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία. Για ποιο λόγο. Για τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων κάνω μια πρόταση που ελπίζω να αποτελέσει και τη βάση της τελικής λύσης. Κατά τη γνώμη μου, η διαφάνεια των αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντική, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου από ανεξάρτητους ε, επιστήμονες. Όμως πρέπει να υπάρχει και ισορροπία στην προσοχή μας και να υπάρχουν ε, διατάξεις που να μπορούν να μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τον τελικό στόχο. Γι' αυτό προτείνω να ορίσουμε τα συνοπτικά αποτελέσματα σε ένα νέο παράρτημα 3α που μετά θα μπορεί να τραποποιείται με πράξεις καταξιοδότηση που σε γενικές γραμμές δεν βλέπουμε καθόλου θετικά αλλά εδώ θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική λύση. Από την άλλη υπάρχουν και εναλλακτικέ προτάσεις για τις ε, κλινικές, ε, για τις δημοσιεύσεις κτλ. και τις μορφές που μπορούν να πάρουν οι δημοσιεύσεις αυτές. Εδώ έχω σοβαρές επιφυλάξεις. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα που δημοσιεύονται. Μπορεί να τίθεται θέματα ανταγωνισμού, ε, στην φαρμακοβιομηχανία, χωρίς όμως αυτό να δίνει κάποια ουσιαστική, αν θέλετε, περισσότερη εγγύηση στην αξιοπιστία των δεδομένων. Πιστεύω είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το ζήτημα. Η μεγαλύτερη διαφάνεια από ό,τι ισχύει σήμερα είναι αναγκαία. Αλλά να λάβουμε υπόψη και πώς έχουν τα πράγματα στην πράξη. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μου σχόλια Ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει να φύγω πριν αρχίσουν οι ψηφοφορίες και ζητώ ε, και πάλι να ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, Κρίστιν, για την ε, τρόπο με τον οποίο διχειρίστηκε σε αυτό το φάκελο και τη σκληρή δουλειά που έκανε με τους κοιόδε. Ο Φιλίν Σουβάν έχει το λόγο να μας πει για τις ε, τροπολογίες του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επενθυμίσω ότι το κείμενο της Επιτροπής είναι πολύ καλό. Θεωρώ ότι θα βελτιώσει πραγματικά την κατάσταση ε, στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τι κλινικέ δοκιμέ, παρότι θα μπορούσαμε και πάλι να επιφέρουμε περαιτέρω βελτιώσει στι προτάσει τη Επιτροπή. Ε, και οι προτάσει του συγγητή προ αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τον συγχαίρω. Σε δύο σημεία θα ήθελα να αναφερθώ για όλες τις ε, τροπολογίες που έχω καταθέσει. Το πρώτο αφορά αυτή τη διάταξη που έχει εφαρμόσει η Επιτροπή, δηλαδή να υπάρξει διάκριση από εδώ και πέρα ε, ανάμεσα στις κλινικές δοκιμές, ε, ανάμεσα σε αυτές που είναι low intervention και στις υπόλοιπες. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να μιλάμε για low intervention, αλλά για low risk, χαμηλού κινδύνου κλινικές δοκιμές λοιπόν. Και δεύτερον, διαρωτώ κατά πόσο είναι σκόπιμο να διατηρήσουμε δύο κατηγορίες αντί για περισσότερες. Κάτι που αυτή τη στιγμή κάνει ο ΩΣΑ και αρκετές χώρες ε, μέλη του ΩΣΑ ε, ε, κινδυνεύουν να έχουν διαφορετικά συστήματα ουσιαστικά. Μετά, σε ό,τι τη διαφάνεια δεδομένων, είναι από πολιτική άποψη σημαντικό ζήτημα και δεν μπορούμε να το χειριστούμε από ιδεολογική σκοπιά. Δύο ζητήματα δεν πρέπει να τα συγχαίουμε. Πρώτον, πρέπει, όπω είπε η Επιτροπή, τα αποτελέσματα, τα πορίσματα των μελετών αυτών να δημοσιεύονται και να έχει πρόσβαση σε αυτά σε όλου. Να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά. Όμω εδώ πέρα δεν μιλάμε για όλα τα δεδομένα. Για τα προσωπικά δεδομένα που δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευση βεβαίω. Είναι δύσκολο να κάνει κανένας οτιδήποτε με αυτά. Μιλάμε για ε, ολοκληρωμένα συνολικά στοιχεία για να μην ε, υπάρχουν ε, παρανοήσεις. Αυτός ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας θα πρέπει όμως να ορίζεται. Αυτό το σύνολο πρέπει να είναι ένα σύνολο που έχει αναλυθεί. Αλλιώς αυτό δεν έχει συμφέρον για το κοινό. Ε, ας πούμε στον ιστότοπο του FDA, ε, τον είπα, μπορείτε να δείτε αυτά τα απορίσματα με πολύ παιδαγωγικό και ενδιαφέροντα τρόπο παρουσιάζονται. Ένα δεύτερο στοιχείο που δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο, είναι ότι όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους όσοι έχουν ε, θέλουν να τα επανυπολογίσουν σε όσους κάνουν περαιτέρω μελέτες. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια διάκριση μεταξύ των δύο. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά. Uh, thank you very much, uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ. Øh, øh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουσόη για το ενδιαφέρον σχέδιο εκθέσεως, γνωμοδοτήσεως μάλλον, πιο σωστά. Και εγώ λίγο πολύ συμφωνώ με τις τροπολογίες του κύριου Μπουσόη. Με απογοητεύουν ωστόσο κάποιες από τις άλλες, όχι του εισηγητού για τους σοσιαλδημοκράτες είναι απαραίτητο, είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Αυτό είναι σημαντικό για τους ασθενείς, αλλά βέβαια και για την κοινή γνώμη συνολικότητα. Όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας των κλινικών ερευνών. Εφόσον βελτιωθεί η διαφάνεια, θα υπάρξει νομίζω και μεγαλύτερη υποστήριξη για ένα μεγαλύτερο αριθμό δηλαδή κλινικών ερευνών, το οποίο είναι απαραίτητο για την ε, προστασία της δημόσιας υγείας. Άρα πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα αποτελεσματικό, μη γραφειοκρατικό σύστημα από τη μια μεριά για τις κλινικές έρευνες και από την άλλη μεριά για ε, υψηλή προστασία των ασθενών. Αυτό είναι το κλειδί, η διαφάνεια. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Ίσως να μην το ανοίξουμε εντελώς για τα λεγόμενα raw data, ακατέργαστα δεδομένα δηλαδή. Νομίζω ότι είναι αυτό το σωστό βήμα. Η ομάδα των σοσιαλδημοκρατών δηλαδή αυτή την ιδέα θα προωθήσει, σας το λέω ήδη, από τώρα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξεύρουμε σωστή λύση με την συνεργασία. Um, ähm, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την καλή δουλειά που έκανε, λέει η κυρία Ρούλε. Θα συμφωνήσω με την κυρία Σουαλδιωμός Στη Γερμανία διεξήχθη συζήτηση, δημοσίως δηλαδή, που περιέλαβε και ορισμένε ανησυχίε. Ανησυχίε δηλαδή ότι υπονομεύεται η ασφάλεια των προσώπων που συμμετέχουν στις έρευνες αυτές. Και διαφάνεια πρέπει να υπάρχει και υπέρ αυτών, εφόσον δηλαδή γίνονται έρευνες επί των προσώπων αυτών, πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Γιατί αλλιώς προκαλούμε φόβους, ανησυχίες που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλη τη διαδικασία. Άρα, επ' αυτού πρέπει να καταλήξουμε οπωσδήποτε σε καλές συμβαστικές προτάσεις. Και εσείς είσαστε εδώ εκ μέρους της κυρίας Μακλάρκιν. Άλλος κανείς, πριν δώσω το λόγο στον Άλαν Μπιέλαν, έχετε το λόγο. Ναι, εγώ μιλώ εξ ονόματος της Έμα Μακλάρκιν, συναδέλφου μου στην ομάδα των συντηρητικών και με παρακάλεσε να σας επισημάνω ορισμένες τροπολογίες, 20 περίπου που κατέθεσε, με στόχο να ξεκαθαριστούν ορισμένες πτυχές ε, του προτινόμενου κανονισμού. Πρώτον, ο ορισμός του Reporting Member State – που πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε ένα, μια χώρα μέλος και σε πλήρες χώρες μέλη όταν ε, συνεργάζονται αλλά κάνουν μια εκτίμηση. Όταν έχει εγκριθεί μια σειρά ερευνών σε μια χώρα μέλος και πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλες, πρέπει να τεθεί το ερώτημα εάν η άποψη της μιας χώρας μέλους εκπροσωπεί άποψη γενικά της Ένωσης. Γι' αυτό έχει υποβάλει τροπολογίες για να ε, ξεκαθαριστεί αυτό καθώς και το θέμα του reporting member state. Προτείνει επίσης τροπολογίες στο άρθρο 6 για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε η reporting member state να κάνει μια πρώτη αξιολόγηση και ότι υπάρχει και αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των ε, δεδομένων. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι προκειμένου είναι να αποφύγουμε μια ενδεχόμενη κατάσταση όπου ενδιαφερόμενη χώρα μέλος θα υποβάλει σχόλια την reporting member state μέχρι την τελευταία ημέρα της ε, περίοδου αξιολογήσεως όπου θα πρέπει δηλαδή να υποβληθεί η έκθεση στους ε, sponsors και στις άλλες χώρες μέλη. Και για το άρθρο 6 πάλι επίσης προτείνει να διατηρηθεί η ισχύουσα διάταξη με μακρότερες προθεσμίες για τις εισρωές των εμπειρογνωμόνων. Όταν πρόκειται για θεραπευτικά ιατρικά ε, προϊόντα ιδιαίτερα προωθημένα. Και είναι δυνατόν αυτό να γίνει υπό την ισχύ τη παρούσα οδηγία και για τι περιπτώσει αυτέ η κυρία Μακράρκιν θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί. Στο άρθρο 9 η κυρία Μακράρκιν θεωρεί ότι η κρίση ανεξάρτητης Επιτροπής Διοντολογίας πρέπει να είναι σαφώς καλυμμένη από την πρόταση και επομένως να αναφέρεται ρητά. Στο άρθρο 39 επιθυμεί να ξεκαθαριστεί η υποχρέωση των ε, χορηγών για, τις, ε, για την υποβολή ετησίων εκθέσεων. Τέλος, θα ήθελε ο κανονισμός να εφαρμόζεται πλήρως. Good. thank you very much. Uh, Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να παρέμβει. Πριν ε, δώσουμε το λόγο στον Θεόφανο Όρος, να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση ότι δεν ε, θα υπάρξει, ε, δεν θα σερβιριστεί καφές εντός της αιθούσης, υπάρχει όμως έξω η αντίστοιχη υποδομή. Καταλαβαίνω βέβαια το πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ και εγώ να πάρω θέση εν μέσω απεργίας, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Μπορείτε να βρείτε καφέ λοιπόν έξω. Και πάλι υπενθυμίζω, σας παρακαλώ να έχετε τις ε, κάρτες σας ε, μαζί σας πριν την ψηφοφορία, γιατί πρέπει να ελέγξουμε τους αριθμούς. Στέφανα Σόρος, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο κύριος Μπούσόη για μένα μπορεί να τρέξει κατευθείαν στο αεροδρόμιο, γιατί συμφωνούμε απολύτως με τα όσα είπε. Δεν ε, έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε. Να, να μείνει απλή διαδικασία. Ε, να μείνουμε ανοιχτοί σε ό,τι αφορά το opt-out, την ε, Επιτροπή Ιδαντολογίας για την πλήρη συνένεση. Θα αναφερθούμε κυρίως στις παρεμβάσεις ορισμένων σκιωδών. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσει. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την προστασία των υποκειμένων, ισχυριζόμαστε έντονα ότι δεν μειώνεται το επίπεδο προστασία των υποκειμένων σε σχέση με την οδηγία που, έχει, που βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγμή και για τη διαφάνεια. Και πάλι να υπογραμμίσω ότι εδώ μιλούμε για δύο πράγματα. Πρώτο και σημαντικό, η διαφάνεια και η δημοσίευση δεδομένων που αφορούν ε, σκευάσματα που έχουν τεθεί υπό αδειοδότηση για θέσεις αγορά. Αυτό δεν έχει σχέση με την νομοθετική πρόταση έχει κάποιε επιπτώσεις και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά έχει σχέση με την ρύθμιση ε, της για τη θέση σε εμπορία. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη δημοσιότητα των δεδομένων. Ε, τώρα, για το σχέδιο κανονισμού που ρυθμίζει εν γέννη τις κλινικές δοκιμές, όλες τις κλινικές δοκιμές δηλαδή και τις μη εμπορικές, Δηλαδή όχι από τις μεγάλες ε, φαρμακευτικές, αλλά από μικρά ιδρύματα, από δημόσια πανεπιστήμια. Εκεί πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο προσεκτικοί, να μην τους επιβάλλουμε ε, δυσανάλογα και παράλογα βάρη. Εάν υπάρχουν ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις στην δική σας εκλογική περιφέρεια, να τις επισκεφτείτε αν υπάρχει ας πούμε, κάποιο μικρό νοσοκομείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πάλι να πω ότι θα εξετάσουμε τις προτάσεις του κυρίου Μπουσόη και εφόσον πρέπει να τρέξει να πάρει και το αεροπλάνο του θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ναι, έφυγε πράγματι ο κ. Μπουσόη για το συνέδριο του κόμματός του, αλλά άκουσε τα όσα είχατε να πείτε. Κυρία Πέρα, συγγνώμη, δεν σας είδα προηγουμένω. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, παρακαλώ. Euh, euh, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την πλειονότητα των επιχειρημάτων του κ. Ζουβάν. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε ό,τι αφορά την ε, προώθηση και ενίσχυση της διαφάνειας. Ε, είναι κάτι το οποίο συζητούμε γιατί πράγματι είναι πολύ καλή η διαφάνεια, αλλά μέχρι πού πρέπει να φτάνει αυτή. Συμφωνώ εδώ με την Επιτροπή που μιλά για μια ποικιλομορφία των ε, κλινικών δοκιμών. Με αποτέλεσμα να μην είναι τις ίδιες εμβέλειας όλες οι δοκιμέ και ούτε να περιλαμβάνουν τα ίδια δεδομένα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πιστέψω την προσοχή σας στο γεγονό ότι η απόλυτη ολοκληρωτική διαφάνεια κάποιες φορές μπορεί να είναι αντιπαραγωγική. Και εδώ θα αναφέρομαι και στο επιχείρημα του κ. Ζουβάν που είπε ότι αν δημοσιεύσουμε τα ακατέργαστα ή μεμονωμένα δεδομένα των επιμέρους προσώπων δηλαδή, μπορούμε να δημιουργήσουμε σύγχυση στο κοινό, που βεβαίως ακριβώς για λόγους διαφάνειας θα ψάξει αυτές τις πληροφορίες, όμως αυτές θα είναι δυσνόητες, δυσανάγνωστες και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και προβληματισμό μάλλον στο κοινό. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Από την άλλη, τα δεδομένα που έχουν αναλυθεί έχουν τύχη επεξεργασία και παρουσιάζονται με, τεκμηριωμένα επιχειρήματα που θα επιτρέψει στο κοινό ή ε, στους ασθενείς, ε, τους ενδιαφέρουμενους ασθενείς να το εξετάσουν, εκεί βεβαίως δεν έχουμε πρόβλημα. Ε, βέβαια έχουμε και κλινικές δοκιμές που αφορούν την αξιολόγηση ε, φαρμάκων και οι ιδιοκτήτες είναι και οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών δεδομένων, προσωπικών δεδομένων. Εκεί λοιπόν υπάρχει και θέμα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια ισορροπία. Ένα ερώτημα που έχω αφορά την διεύρυνση των μελετών σε άλλα κράτη-μέλη. Για μένα εξακολουθεί να υπάρχει μια σύγχυση. Θα ήθελα να έχω κάποιες διευκρινήσεις από αυτού. Σε ποιο πλαίσιο λοιπόν ε, επιτρέπουμε τη διεύρυνση σε νέα ερευνητικά κέντρα, θεωρώ σκόπιμο όταν υπάρχει μια κλινική δοκιμή που έχει λάβει ε, έγκριση, αδειοδότηση, αλλά δεν μπορεί ας πούμε το ερευνητικό κέντρο να βρει τον απαραίτητο αριθμό ασθενών, τότε πράγματι μπορούμε να κοιτάξουμε σε άλλα κρατημέλη, αρκεί βεβαίως να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη αυτού του κράτους μέλους σε ό,τι αφορά τα αντιοντολογικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Well, since we have a bit of time before the vote, uh, if Έχουμε λίγη ώρα ακόμα ε, πριν από την ψηφοφορία. Στέφανο, θες να απαντήσεις μήπως? Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Θα μιλήσω στα γαλλικά, καθώς ε, στα γαλλικά έγινε παρατήρηση. Υπάρχει μια διαδικασία που προβλέπεται για την ε, επέκταση σε νέα ερευνητικά κέντρα και νέα κράτη-μέλη, όμως ε, αυτή βασίζεται στην διαδικασία της ε, έγκρισης, της συνένεσης. Μόνο το δεύτερο τμήμα του φακέλου, λοιπόν, που υποβάλλεται στις ε, αρχές, υπόκειται σε επιπλέον αξιολόγηση για ένα νέο κέντρο ή ένα νέο κράτος μέλος. Επίσης, στηρίζω τα όσα υπόθηκαν για τη διαφάνεια Πολύ σύντομα θα ήθελα να επισημάνω ότι οτιδήποτε συνδέεται με την ε, διάχυση δεδομένων κλινικών δοκιμών για, την, ε, για διοδοτημένα φάρμακα διαφέρουν από τη διαφάνεια στις κλινικές δοκιμές που συνδέονται ε, που συνδέονται με τη σύγκριση με υφιστάμενα φάρμακα από ερευνητικά κέντρα, από δημόσιε αρχέ ή από φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αναφερθήκατε λοιπόν στη διαφάνεια, γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω όσου θα εξετάσουν αυτό το κείμενο να λάβουν υπόψη και το διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για, την, ε, για, για τα δεδομένα αυτών των κλινικών δοκιμών. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ο εισηγητή ε, έπρεπε να φύγει, επομένω προφανώ δεν μπορεί να πάρει το λόγο κλείνοντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Να ευχαριστήσω λοιπόν ε, τον Κρίστιαν, ε, παρότι δεν είναι εδώ μαζί μα. Να ευχαριστήσω και του σκιώδει και για τι συμβιβαστικέ. Το χρονοδιάγραμμα. Θα τις εξετάσουμε στις 20 ε, Μαρτίου τις συμβαστικές. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ε, την 21η Μαρτίου και στη Λίμπε στις 24 και 25 Απριλίου. Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, ακόμα καταφθάνουν οι συνάδελφοι, να σας ε, καλωσορίσω λοιπόν. να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και ένα νέο ε, ενημερωτικό φυλάδιο, το οποίο μπορείτε να λάβετε. Δεύτερον, στα πρακτικά ζητήματα. Επαναλαμβάνω ότι δεν ε, θα σερβιριστεί καφέ ε, μέσα στην αίθουσα σήμερα, όμως μπορείτε να βρείτε καφέ έξω. Αν θέλετε λοιπόν καφέ πριν ξεκινήσουμε. Όπω υπόθηκε και στην ακρόαση χθε, είναι μια υπηρεσία που αυξάνει την παραγωγικότητα. Δεν ε, θα μα ε, παρασκευθεί λοιπόν μέσα στην αίθουσα, μπορείτε να βρείτε όμω καφέ έξω. Και τέλο, παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί την ε, κάρτα σα, γιατί υπάρχουν κάποιε ψηφοφορίε όπου θα πρέπει να ελέγξουμε του αριθμού. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Right. Um, I'm going now to move on to the uh, votes. τώρα στις ε, ψηφοφορίες που έχουμε για σήμερα το πρωί. Έχουμε μία σειρά ψηφοφοριών που οι και οι σκιώδες ζητούν εντολή από την Επιτροπή για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ώστε να υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Για αυτούς τους φακέλους καλώ τους ηγητές να σας το δηλώσουν και μετά θα ψηφίσουμε χωριστά. Να σας υπενθυμίσω ότι βάσει του κανονισμού για να διασφαλιστεί η εντολή πάνω από το ίμιση των μελών της Επιτροπής πρέπει να υπερψηφίσουν την πρόταση. Χρειαζόμαστε λοιπόν 21 ψήφους υπέρ για να μπορεί να υπάρξει εγγύηση αυτή τη εντολής. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Λοιπόν, πρώτη περίπτωση. Οδηγία που τροποποιεί την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. Θα καλέσουμε την εισηγήτρια να μας παρουσιάσει την προτασία και μετά πάμε κατευθείαν στην ψήφο. Κύριε Βερνιού. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes. Καλημέρα και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομη παρουσίαση διότι κυρίως επιθυμώ να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους στον φάκελο αυτό. Έχουμε εργαστεί από καιρό στην ομάδα εργασίας που είχαμε ιδρύσει για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και μάλιστα πέρσι, σε συνεργασία με την Κομισιόν, προβήκαμε σε τακτικές συναντήσεις και με όλες, όλους σχεδόν τους και οδησηγητές όλων των πολιτικών ομάδων που καθένας ή καθεμία από αυτούς συνεισέφεραν σημαντικά και βεβαίως και μέσα από τα πλαίσια των διαφόρων παραδόσεων και διαφορετικών νοοτροπιών καταφέραμε μέσω της ΣΥΜΚΟ να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Κοινοβουλίου, όχι μόνο απέναντι στο Συμβούλιο με το οποίο προχωρούμε τώρα σε διαπραγματεύσεις προς το συμφέρον βέβαια των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουμε μέσω της ψηφοφορίας όφελος σε όλες και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδίω, και το τονίζω αυτό, εγώ δεν είμαι οπαδός των συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση, το γνωρίζετε αυτό, αλλά σε αυτό το θέμα πρέπει να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν μακρύτερα αλλά και ω το δυνατόν ταχύτερα. Α μην λησμονούμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια νεαροί άνεργοι στην Ευρώπη για του οποίου η κινητικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη για να μπορέσουν να βρουν θέση στο επαγγελματικό μέλλον. Στην, θητεία, στην, συγγνώμη, στην εντολή αυτή που ελπίζω θα μου δώσετε σήμερα για να διαπραγματευτώ με το Συμβούλιο, το έχω αυτό στο μυαλό μου διαρκώ. Εκτό από το κοινό πλαίσιο εκπαιδεύσεω, εκτό από τι πρακτικέ εκπαιδεύσει στάζ, και μια ε, και επίσης και την επαγγελματική ταυτότητα η οποία θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, εργασίας των επαγγελματιών και των πολιτών μέσα σε πλαίσια ασφάλειας και εμπιστοσύνη. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας λοιπόν και δεσμεύομαι προσωπικά να πράξω τα πάντα σε πλήρη διαφάνεια. Η Ιρλανδική Προεδρία είναι επίσης ενθουσιώδης στο θέμα αυτό και μάλιστα ε, σκέπτεται ας πούμε και στο δικό μας μήκος κύματος. Ευχαριστώ λοιπόν που ε, ελπίζω ότι θα μου δώσετε την σχετική εντολή. Ευχαριστούμε για αυτήν τόσο καλή παρουσίαση. Παρακαλώ, επειδή είναι πολύ σημαντικέ πληροφορίε, θέλω να κάνω και κάποια γενικά σχόλια που αφορούν όλε αυτέ τι συμφωνίε που συζητήσαμε με του συντονιστέ και του συζητητέ και του κοιόδη μάλιστα προβλέπεται σε κάθε συναντή τη Επιτροπή πλέον, όταν υπάρχουν τέτοιε προτάσει για το λέει, έτσι δεν θέλω να προδικάσω τα πράγματα, αλλά θα υπάρχει πλέον χώρο, χρόνο στου ηγητέ να παρουσιάσουν την πρώτη διαπραγματεύσεων, τα εκκρεμή ζητήματα και όσα θέλει να μοιραστεί μαζί μα δημοσίω. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο και ελπίζω πραγματικά να αποτελέσει η Επιτροπή μα το παράδειγμα για το πώ γίνονται διαπραγματεύσει στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου θα, στους διαλόγου, διαλόγους εγώ θα προείσταμαι πάντοτε, θα είναι παρόντες βεβαίως ο συζητητής και σκιώδες. Και αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Οπότε από τα μέσα Απριλίου και μετά θα είμαστε πραγματικά πάρα πάρα πολύ α, βαρημένοι. Ο κύριος Σφαν ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τα όσα είπατε για τον τριμερή διάλογο. Μεταξύ των συντονιστών εχθές συζητήσαμε και είπαμε ότι επιθυμούμε να διατηρήσουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε ψηφοφορία στην Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού εφόσον το Συμβούλιο δεν κινηθεί προ την δική μα κατεύθυνση. Ναι, είναι θέμα του πώ θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τι διαπραγματεύσει. Ξέρετε, έως σήμερα εγώ δεν έχω δει καμιά τέτοια διάθεση του Συμβούλιο. Αν μα ακούει τώρα η Ελληνική Προεδρία και κάνει τέτοιο σημάδι, να το δούμε. Στη δική σα περίπτωση, στα δικαιώματα καταναλωτών, πράγματι είχαμε κάποιε δυσκολίε. Πήγαμε την ψήφο στην ε, Ολομέλεια και μετά επιστρέψαμε στην Επιτροπή για περαιτέρω Εξετάξεων. Είναι και αυτό, είναι και αυτό πάντοτε μία περίπτωση και μια δυνατότητα που μπορεί πάντοτε ε, να επικαλεστούμε. Με έναν φορτηγό κάπως πυρηνικού χαρακτήρα, αν θέλουμε δηλαδή να απασφαλίσουμε αυτή τη χειροβομβίδα ή όχι, είναι στα διαπραγματευτικά μας, αν θέλετε, ατού. Λοιπόν, τώρα να θέσουμε στην ψηφοφορία την έγκριση της εντολής για να διαπραγματευτούμε το θέμα αυτό. Άρχεται ψηφοφορία. Μπορείτε ε, πραγματικά να επιταχύνετε. Λοιπόν, σιγά σιγά ανεβαίνουμε στου τέσσερις ψήφου. Υπάρχει κόσμο που δεν ψηφίζει. 33. Ποιο θέλει να ψηφίσει. Πέρας ψήφου. Εγκρινέται με 28 ψήφους υπέρ, 4 κατά και ε, δύο Ξεκάθαρη η εντολή, κάθε επιτυχία σε ευχόμαστε. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση της κυρίας Λεγκρίπ. Εδώ είσαστε, αλλά είσαστε πίσω. Ε, κάθεστε πίσω, μάλιστα. Θα πάρετε το λόγο για τον ενωσιακό τηλεμιακό κώδικα, κυρία Λεγκρίπ. Η κυρία Λεγκρίπ έχει να μας πει πέρα από την εντολή και κάποια άλλα πράγματα για τα οποία θέλει μία έγκριση. Παρακαλώ. Oui, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε λίγο θα ψηφίσουμε για την εντολή που θα μπορούσε να, δοθεί, να δώσει στην ομάδα μας να ε, υπησέλθει σε συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ακριβώς για τον τελωνιακό κώδικα της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή όλες οι πολιτικές ομάδες είναι υπέρ της ε, ανάθεσης αυτής της εντολής διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να επιβεβαιωθεί αυτή η σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών ομάδων. Να διευκρινίσω μόνο το εξή πριν ψηφίσουμε, ε, ο εισηγητή και οι σκιώδη θέλουν να κάνουν μια δήλωση ε, επί της οποίας συμφωνούμε και η οποία θα αναφερθεί ε, και στα πρακτικά της ε, συνεδρίασής Θα σας διαβάσω λοιπόν. Η, εισηγήτρια και οι σκιώδεις εισηγητές συμφωνούν ε, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να Υποβάλλει το Μάρτιο μια τρόπαση, πρόταση τροποποίησης ε, του κανονισμού 4508 του Ελληνικού Κώδικα σε ό,τι αφορά την ημερομηνία εφαρμογής ε, και στο άρθρο 148 παράγραφος 2. Στην περίπτωση όπου οι εξελίξεις των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο δεν θα επιτρέπουν την σύναψη ικανοποιητικής συμφωνίας μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Αυτή η δήλωση, και θα κλείσω εδώ κύριε Πρόεδρε, ε, απευθύνεται δύο, σε δύο σημεία. Πρώτον, εκφράζουμε την πραγματική μας βούληση να διεξαγάγουμε επικοδομητικές και αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε ε, σε αυτή την μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, ε, χάρη σε μια καλή συμφωνία διαπραγματευτική. Και δεύτερον, υπάρχει ένας προβληματισμός σε ό,τι αφορά την τήρηση των ε, δικαιωμάτων μας ως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή ότι εμείς συμμετέχουμε ε, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις βεβαίως με κάθε καλή διάθεση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε την εντολή για τον ενωσιακό, τον κώδικα, αναδιατύπωση και ισχύουν όσα είχα πει και νωρίτερα και εδώ άρχεται η ψηφοφορία για την εντολή μαζί με την δήλωση της κυρίας Λεγκρίπ. Πέραση ψηφοφορίας. 35 ψήφοι υπέρ και μία ψήφος κατά, ξεκάθαρη εντολή και πραγματικά προσβλέπουμε στην επιτυχία της προσπάθειάς σας. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση για τις αναθέσεις συμβάσεων παραχώρησης. Ο κύριος Φιλίπ Ζουβάνο έχει το λόγο. Euh, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μας δώσετε εντολή και ε, για το ζήτημα των ε, συμβάσεων παραχώρησης, ε, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και ένα χρόνο τώρα. Υπήρξε μεγάλη ε, πλειοψηφία σε όλα τα κόμματα ε, στην ψηφοφορία. Γι' αυτό και μπορούμε να πάμε σε αυτόν τον τριμερή διάλογο. Ε, αρκετά ζητήματα έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο και αυτές οι εξελίξεις μάλλον αυτές, αυτά τα στοιχεία που την χάνουν ευρεία συνένεση θα τα παρουσιάσουμε στον τριμερή διάλογο. να προσθέσω ότι η ομάδα διαπραγμάτευση θα εξακολουθήσει να είναι εξαιρετικά προσεκτική ε, κατά την προσπάθεια εξέβρεσης ε, εξισορροπημένων ε, λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ιστορικά παραδοσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητε μας και να πω στους Γερμανούς και Αυστριακούς συναδέλφους που αυτή τη στιγμή έχουν έναν εξαιρετικά πολιτισμένο βέβαια διάλογο, γιατί έχουμε και εκλογές στη Γερμανία, ότι ε, εμείς ε, παρακολουθούμε τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως και ο Επίτροπος Βαγνιέ. Ο Επίτροπος Βαγνιέ που θα έρθει στην Επιτροπή μας ε, στη συνέχεια θα εκφράσει και τη βούλησή του να βρει νέες λύσεις και να εξελίξει το κείμενο προς μια κατεύθυνση που θα είναι από πολιτική άποψη ικανοποιητική για όλους. Κατά τη γνώμη μας υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης για να επιφέρουμε πραγματικά σημαντικές βελτιώσεις. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much, uh, um, Καλώς, λοιπόν. Ας περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Φιλίππ. Νομίζω ότι είχες και κάτι να μας διαβάσεις για την εντολή. Όχι. Σας διάβασα μια πρόταση που για μένα ήταν εξαιρετικά σημαντική, που διευκρινίζει ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης θα εξακολουθήσει να ε, προσπαθεί την, να εξεύρει την, μια ισορροπία για στοιχεία τέτοια ιστορικά που χαρακτηρίζουν αυτούς τους κλαδικούς τομείς και όλα αυτά τα στοιχεία η ομάδα διαπραγμάτευση σα διαβεβαιώ ότι θα τα υποστηρίξει κατά τις... τον τριμερή διάλογο. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό είναι το, κύριο. Uh, the vote then is... Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία ώστε η διαπραγματευτική ομάδα να πάρει εντολή για να αρχίσει διαπραγματεύσει για την πρόταση που αφορά τη συμβάση παραχώρηση. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 25 ψήφου υπέρ, 10 κατά και δύο εποχέ. Καταφέραμε λοιπόν να ξεπεράσουμε το σημείο αναγκαίε ψήφους και περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθούν οι συζητήσεις. Σας υπενθυμίσω ότι όλοι οι συγητές θα έχουν πλέον το χρόνο στι συνεδριάσει τη Επιτροπή μα για να μα ενημερώνουν για το πώ προχωρούν οι διαπραγματεύσει. Πάμε τώρα στι δύο τελευταίε προτάσει και προτείνω να δούμε από κοινού τι δύο προτάσει ε, ταραμπέλαν και είναι δύο διαφορετικές ε, οδηγίες. Δημόσιες συμβάσεις ως κλασική οδηγία και οι δημόσιες συμβάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες κυρίως ωφελίας, ύδατος, ενέργειας, μεταφορών κτλ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ταραπέλα να μας παρουσιάσει και τις δύο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να μας δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια εντολή διαπραγμάτευσης ε, με το Συμβούλιο μετά την ε, τελευταία συνεδρίαση με τους Κιώδης ε, καταλήξαμε σε τρία αιτήματα. Έτοιμα για αξιολόγηση αντικτύπου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την ΚΟΕ αλλά και από την Άλντε. Βεβαίως, αυτό αφορά οποιαδήποτε προθεσμία για αυτή την ομοδότηση. Ω εισηγητή, ε, θεώρησε σημαντικό να αναφερθεί και στην Επιτροπή μας ε, η εξέλιξη των ε, συζητήσεων στον τριμερή διάλογο, τα ζητήματα που έχουν προοδεύσει, τα ζητήματα που είμαστε στάσιμοι, σε ό,τι φορά τη διαφάνεια, ζητήματα που έχουν παρουσιαστεί και έχουν συζητηθεί και μεταξύ σκιωδών και με εσά, ε, κύριε Πρόεδρε, αλλά και με επαφέ που είχα στην ε, Επιτροπή και στο Συμβούλιο με την ε, Ιρλανδική Προεδρία. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρηθεί αυτή η διαφάνεια. Τρίτον, θεωρώ ότι υπάρχει ένας πολύ σημαντικός δεσμός και σύνδεση μεταξύ των δημοσίων προμηθειών και των παραχωρήσεων, των συμβάσεων παραχώρησης. Είναι Καλό λοιπόν να μείνει αυτός ο παραλληλισμός μεταξύ των δύο θεμάτων και μάλιστα να πω ότι και εκεί υπήρχε ευρεία συνένεση και πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Συμβαστικές προτάσεις τυχάνουν ευρεία συνένεση λοιπόν. Άλλες όχι, ίσως για λόγους κατανόησης θεωρώ που βεβαίως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μπορεί να βρεθεί πάλι μια συμβαστική λύση. Ελπίζω λοιπόν να λάβω την εντολή από εσάς. Ευχαριστώ. Well, thank Ευχαριστούμε θερμά και ευχαριστούμε και για τον ηγετικό σας ρόλο. Όπως ε, αυτό φορά και όλους οι ηγητές, γιατί πραγματικά είναι περίπλοκο αυτό το θέμα. Να σας πω ότι για να μπορέσει αυτή η οδηγία να γίνει φιλική για τις μικρές επιχειρήσεις που είναι και αυτό που επιθυμείτε όλοι σα και όσοι μας ακούτε και μας παρακολουθείτε αυτό επιθυμείτε, αυτό είναι ο στόχος μας. Λοιπόν, αυτή την εντολή τη θέτουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ή μάλλον ξεκινούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένα παραπάνω μέλο του ΕΛΚ, παρακαλώ, κάποιο να βγάλει την κάρτα. 31 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά, ξεκάθαρη εντολή. Καλή τύχη λοιπόν σε όλου του ηγητέ. Είπαμε ότι θα τα παρακολουθούμε τα θέματά σα πολύ στενά. Πιστεύω ότι σημαίνει ότι θα έχουμε περιμένει ατζέντα, αλλά θα μα επιτρέπει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Προχωρούμε τώρα σε μια σημαντική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση τη κυρία Τούρνεν για την ε, ε, επιτροσία στην αρμόδια επιτροπή απασχόληση. Αφορά την απόσπαση εργαζομένων. Θέλει να πει λίγα λόγια η συγγήτρια. Ναι, εντάχει. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους κοιόδης. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσαν και σκληρή τροπορτινά άσκηση, όμως πολύ σημαντική να γίνει. Στόχο στόχος είναι μια ισχυρή ιστορική αγορά με το κατάλληλο επίπεδο προστασίας για τους εργαζόμενους, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά στοιχεία που τόσο συχνά βλέπουμε με την κατάχρηση ε, που γίνεται στους εργαζομένους με χαμηλούς μισθούς και ταυτόχρονα διαδικασίες να είναι εύκολες και διαφανείς για τις επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στο εξωτερικό. Καταφέραμε να έχουμε συμβιβαστική λύσεις λύσει για όλε και τον άρθρα με του κοιόδε. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο επίτευγμα και θα πρέπει να το επισημάνω. Βεβαίω υπάρχουν κάποια άρθρα στα οποία δεν υπάρχει συμφωνία και πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για τη σκληρή δουλειά και το δικό μου προσωπικό που τους οφείλω τα μάλλα. Ωραία, λέει ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Πραγματικά κάνετε σκληρή δουλειά για να καταφέρετε μια συμφωνία. Είναι ε, δεδομένο όμω ότι υπάρχουν και κάποιε διαφωνίε. Θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, γιατί σε κάποια σημεία θα είναι μάλλον α, δύσκολο να βγάλουμε αλλιώ το συμπέρασμα. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε γρήγορα, γιατί 10 και 4 θα έχουμε τον Επίτροπο πιστεύω θα κλείσουμε έως τότε, αλλά παρακαλώ να είστε γρήγοροι. Οι κύριοι Κέχαρτ και Σουάπ να μου δείξουν. Ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ. Πρώτο, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, εκκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 1, τμήμα 2 λοιπόν, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα Τροπολογία 189 του κυρίου Τιγιόν. Λοιπόν, τροπολογία 189. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία συμβιβαστική 2 υπέρκατα, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 181. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάω τώρα στην τροπολογία της συμβαστική 2α. Άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στο 194. 194 άρχεται ψηφοφορία. Ε, απορρίπτεται. 195 του της εισηγητρίας άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 54 αποσύρεται. 196 άρχισε φοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στη βαστική τροπολογία του όπου χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται ξεκάθαρα. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται ξεκάθαρα και αυτό. Οπότε πάμε στην τροπολογία 55 που είναι αρκετέ σελίδε πιο κάτω. Σελίδα 10. Μπράβο, πολύ καλή δουλειά κάνατε, κύριε Τεθέλ. Λοιπόν, τροπολογία 55 της εισηγήτριας, υπέρ, κατά εγκρίνεται. και τροπολογία του άρθρου 5. Υπερκάτα. κατά. Πάμε τώρα στη σελίδα, 200, σελίδα 12, τροπολογία 243. Υπέρ. Να το κοιτάξουμε. Παρακαλώ, έρχεται η ψηφοφορία. Το ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 ψήφους υπέρ και 17 κατά. Συμβαστική για το άρθρο 6 υπέρ κατά. Εκρίνεται. Άρα πάμε στη συμβαστική για το άρθρο 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη τροπολογία 77 της εισηγήτριας. Υπέρ. Ας το δούμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Λοιπόν, η τροπολογία 77 της εισηγήτριας. και τη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ 15 κατά τροπολογία 78 της εισηγήτριας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 9 υπέρ. Και εδώ πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία το άρθρο 9. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα πρέπει να δούμε όλες τις τροπολογίες. Υπομονή. Η 261 αποσύρεται. 79 της ηγητρίας. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να την ελέγξουμε και αυτή. Λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για την 79 της εισηγητρίας. Πιστεύω ότι απορρίπτεται, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. Παρακαλώ να είστε γρήγοροι. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. 262. Άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 264. Άρχεται η ψηφοφορία της κυρίας Πετικάινεν, τροπολογία. Απορρίπτεται. 263 αποσύρεται και μετά έχουμε ένα μπλοκ τροπολογίων ε, για διαγραφές του κυρίου ε, Λόκενγκάρτ. 265-274 απορρίπτεται ξεκάθαρα. 266 της κυρίας Χάνσλικ. Υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Είναι σημαντική για αυτή η τροπολογία. 266 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά η 80 της ηγήτριας υπέρ. Και εδώ και πάλι. Ας το δούμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 81 της ηγητρίας. άρχιε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 270 της Χάνσλικ. Άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Θα στη 273. 273 λένε τα χαρτιά μου της κυρίας Χίρς και Κρότσμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά η 83 της συγγήτριας. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οπότε πάμε στη 275 τη κυρία Χάνσλικ και των λοιπόν. Άρχεται ψηφοφορία για το 275. Πέρας. Α, απορρίπτεται. πολύ καθυστερημένος. Εγώ, μόλι ανακοινώ τα αποτελέσματα, ξέρετε, όταν έχουμε ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αλλαγή ψήφου. Τώρα που είμαστε 276. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 276. Προσέξτε τι ψηφίσετε και γρήγορα. Απορρίπτεται. 84 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 277 της ε, κυρίας Τεγιόγκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 85 της εισηγήτριας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 86 της εισηγήτριας. Ψηφίζουμε. Πιο γρήγορα. Πέρας. Απορρίπτεται. 278 του κυρίου Λόκενχαρτ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 87 της συγγετρίας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 279 της κυρίας Γκέπαρτ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 280 της ηγετρίας υπέρ. Ας το δούμε ηλεκτρονικά. Ας το δούμε ηλεκτρονικά. 280 της ηγετρίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 281 αποσύρεται. 283. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 88 της ηγετρίας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 282. Κιουσβάπ. υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και 89 της ηγητρίας. Αρχίζουμε να ψηφίσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα συμβαστική για το άρθρο 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ωραία. Πάμε στο άρθρο 11 σε δύο τμήματα. Τμήμα 1 της συμβαστικής για το 11. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται, ξεκάθαρα. Τμήμα 2. Άρχεται η ψηφοφορία για το τμήμα 2. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στο 294. Μία σειρά τροπολογιών για διαγραφές υπέρ. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θα το ελέγξουμε. Άρχεται ψηφορία ηλεκτρονικά για αυτό το μπλοκ τροπολογιών. Yeah, That's carried. So we now go to, um, Τώρα λοιπόν Α, εκπίπτει η συμβαστική 12 λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Α, μάλιστα, διαγράφεται λοιπόν. Ωραία, λοιπόν συμβαστική 13. Κύριε Τουρίνεν, προκλήθηκε νομίζω κάποια σύγχυση. Ας διευκρινίσω. Εκπίπτει η συμβαστική 12 αφού εγκρίθηκε η 294 Αυτό, αυτό. Επειδή εδώ, γύρω μου υπήρχε κάποια σύγχυση. Η 12 ε, καταπίπτει, δεν, δεν, ε, δεν παίζει πια, λέει ο πρόεδρο, γιατί καταργήθηκε το άρθρο. Ωραία. Τρο, συμβαστική τροπολογία 13, υπέρ. Πρόκειται για ψηφοφορία κατά τμήματα, σε δύο τμήματα. Λοιπόν, τμήμα πρώτο, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κύριε Τούρινεν, νομίζω να επαληθεύσετε, πρόεδρε, για διαδικαστικούς λόγους. Εφόσον ψηφίσουμε τις τροπολογίες, Κοιτάξτε, η ερμηνεία που δίνουμε εδώ και που νομίζω ότι είναι σωστή, είναι περάσαμε όλες τις προτάσεις κατάργησης του άρθρου 12 και όλες τις σχετικές υποπαραγράφους. Άρα δεν υπάρχει πλέον χώρος ε, για τις ε, συμβαστικές γιατί δεν υπάρχει και το άρθρο. Άρα νομίζω ότι η αποφάση ήταν σωστή. Τώρα, για το τμήμα δεύτερο της 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα, Προχωρώ. Στο 108. 108 του εισηγητή. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση δηλαδή. Πέρα ψήφου. Απερίφθη. 109 εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 110 εσύ το υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μια στιγμή. 327. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και αυτή εδώ εγκρίνεται. Άρα εκπίπτει 111. 112. Οι φιλελεύθεροι βλέπω τον κύριο Μάντερ. Ε, δείξτε καθαρά με τον αντίχειρά σα προ τα πάνω προ τα κάτω. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 3.28, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 3.29, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 113, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Τροπολογία, σημαντική τροπολογία 18, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 118 της εισηγήτριας, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 119 και 333 μαζί υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 120 εισηγητρίας υπέρ κατά απορρίπτεται 121 υπέρ κατά απορρίπτεται 334 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 1 Κάτι λέει εδώ για το παραδεκτό, παρόλα αυτά να την ψηφίσουμε. Τροπολογία λοιπόν, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 123 έχει αποσυρθεί, 124 υπέρ. Κατά. Αυτή επίσης απορρίπτεται καθαρά. 125 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 2 αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας απερίφθη αυτή άρα προχωρούμε τώρα στα εκτιμώντας και αρχίζουμε το 127 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 εισηγητρίας υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 129. Handslick υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πολύ κοντά, εν πάση Άρα, η 128 εκπίπτει, η 3 τώρα τη ηγετρίας υπέρ, νομίζω χρειάζεται επαλήθευση. Τροπολογία 3 της ηγετρίας. Πέρας, 20 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. 130 εκπίπτει, 4 της ηγετρίας υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 132 εκπίπτει, 136 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Και ακολουθεί η τροπολογία 6 της συγγήτριας υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 9 εισηγητρίας υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 10 εισηγητρίας υπέρ. Όπως είπα 10 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. 143. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, με συγχωρείτε. Εγκρίνεται, αλλά σε επαληθεύσουμε. Ας παληθεύσουμε. Καλά είναι να κάνουμε και μια επαληθεύση. Εγκρίθηκε, 21-17. 144 υπέρ. Επαλήθευση. Αρχίζει. Πέρασα περίφθη. 19-19. Πάντως κάποιος δεν ψήφισε. 145 και 46 είναι ταυτόσιμες. Αρχίζει. Πέρας. Πάλι ισοψηφία 19-19. 147 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11. Όχι αυτή εκπίπτει καθώς και επόμενη 148. 12 λοιπόν σε ηγητρίες υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14 εισηγήτρια πάντα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 149 De Jong υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 150 Handslick υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται αυτή. Και Προχωρούμε ευθύ αμέσω στην συμβαστική 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά απορρίπτεται. 156 156 ναι. υπέρ κατά εγκρίνεται 157 εδώ κατά τμήματα τμήμα πρώτο, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 17 εισηγητρία υπέρ, κατά. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται επαλήθευση. 17 λοιπόν εισηγητρία. 19 υπέρ 18 κατά. 18 ψηφίζεται 18 υπέρ κατά απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά εγκρίνεται. 159 εισηγήτριες υπέρ κατά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Α, εγκρίνεται σαφώς γιατί το Λαϊκό Κόμμα ψηφίζει υπέρ. 160 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Είναι λίγο λεπτό, λεπτή η κατάσταση εδώ. 162 Αρχίζει. Α, δεν είναι και τόσο κοντά τα αποτελέσματα. Απορρίφθη, σαφώς. 19 της συγκίτριας υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 164. Δε Jong. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 165. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ εγκρίνεται 167 ψηφίζεται καλώς υπέρ κατά απορρίπτεται 20 υπέρ Επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. Με διαφορά δύο ψήφων. Συμβιβαστική επί του εκτιμώντας 23. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ορισμένες τροπολογίες διαγραφής που είναι όλες ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, Εγκρίνονται λοιπόν αυτές οι τροπολογίες διαγραφής, ώστε τώρα προχωρούμε στις άλλες διαγραφές, 23 και επόμενες. 23 και επόμενες λοιπόν, υπέρ, κατά, εγκρίνονται και ακολουθεί 176 υπέρ κατά εγκρίνονται και ακολουθεί Εκατόν Δε De Jong, 180, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω αυτή, αλλά ας το επαληθεύσουμε. για να είμαι σίγουρος. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρασε. Και όντως απερίφθη. 25 εισηγητρία υπέρ. Κατά. Α, η φιλελευθερία είναι υπέρ αυτή τη φορά. Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. 25 αρχίζει η ψηφοφορία. Τρεις δεν ψηφίζουν, άλλος κανείς θέλει να ψηφίσει. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 181. Handslick. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επαλήθευση θέλετε. Καλά. Εγκρίνεται λοιπόν 20, υπέρ 17 κατά. 182 υπέρ κατά. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. 183 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 184 υπέρ κατά. Εγκρίνεται και αυτή. 26 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Όμως αρχίζει η ψηφοφορία παλήθευσης ηλεκτρονική. Πέρας. Απερίφθη. Με μικρή διαφορά. 27. Μεσηγητρίας. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και η 186. Υπέρ. Αρχίζουμε τώρα ψηφοφορία για την 186. Πέρας. Απερίφθη με ισοψηφία. Τώρα, κοιτάξτε, τελική ψηφοφορία αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία, ονομαστική επομένως, πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν με 20 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 4 αποχές. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Τούρνεν. Ήταν όντως δύσκολο το θέμα. Ίσως ορισμένοι, ίσως ορισμένοι παρατηρήσατε ότι δεν υπερψήφισα τελικά το κείμενό μου, διότι περάσαμε ώρες και ώρες και έχουμε καλό προσωπικό. Νομίζω το άρθρο 3 ιδίω είναι ιδιαίτερα ευφυέ. μπορεί λοιπόν να διαβιβαστεί ω γνωμοδότηση, αλλά οφείλω να πω επίση ότι υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα θέματα όπου εγώ απογοητεύτηκα από τι πολιτικέ μα συζητήσει, διότι δεν κατέστη δυνατόν να γίνει ουσιώδης πολιτική συζήτηση για τα άρθρα 9 και 12. Ήταν απόλυτα οχυρωμένες θέσεις και με λυπεί αυτό, διότι Ιδίω για, τα για τα μέτρα ελέγχου του άρθρου 9 έπρεπε να υπάρξει μια πιο ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Είδα και μέλη μακράν των κομματικών τους ε, τοποθετήσεων. Πρέπει να λειτουργήσει όμως την πραγματική ζωή. Για μένα είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Δεν μπορώ λοιπόν να υποστηρίξω πλήρως τη γνωμοδότηση αυτή στην Επιτροπή Απασχολήσεω. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκα να απόσχω το εκφράζω τη λύπη μου, αλλά το δέχομαι. Καμιά φορά κερδίζει κανεί ψηφοφορίε, καμιά φορά χάνει. Ωστόσο δεν μπορώ να υποστηρίξω με την υπογραφή μου τη γνωμοδότηση αυτή. Ελπίζω ότι η πολιτική συζήτηση για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση της απόσπασης των εργαζομένων θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ πάντως και πάλι. Ευχαριστούμε που εκφράσατε τη θέση σας. Ξέρω ότι υπήρξε διαφωνία. Μισό λεπτό είναι σημαντικό. Ησυχία παρακαλώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακριβώς μας είπατε όμως. Είστε ε, ε, σε θέση να μεταφέρετε αυτή την νομοδότησε άλλη επιτροπή ή όχι. Αν έχω την ε, ευκαιρία να βγάλω το όνομά μου από εκεί, θα το ήθελα. Εντάξει, θα προτιμούσα όμως εσείς να το ε, κινήσετε προσωπικά. Ξέρω, κατανοώ τη θέση σας, όμως έχετε καλύτερη γνώση ε, του ζητήματος. Evelyn Gebhardt. I δεν επιθυμώ να βλέπω πρόσωπα να περνούν από τον διάδρομο μπροστά από τα έδρανα των μελών. Όποιος επιθυμεί να αποχωρήσει, το κάνει από τον πίσω διάδρομο. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μου ομάδα ψήφισε ενωμένη κατά της γνωμοδοτήσεως, διότι δεν επιθυμούμε και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε γνωμοδότηση όπου πολύ απλά καταπατούνται τα δικαιώματα των αποσπαζόμενων εργαζόμενων. Ιδίω οι δυνατότητες ελέγχου υπέρ των χωρών μελών για να παρεμποδίζουν την κακή μεταχείριση των εργαζομένων όπως βλέπουμε για παράδειγμα στη Γερμανία να συμβαίνει με την ε, εταιρεία Amazon ο τρόπος που μεταχειρίζεται τις και τους εργαζόμενους και σε άλλες χώρες αλλά και όχι μόνο η Amazon πρέπει να επιτρέψουμε, πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία, τα μέσα στις αρχές μας να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Και εδώ αυτό που προτείνεται είναι να μείνουμε και πιο πίσω και από τα όσα περιλαμβάνει η ε, οδηγία για την απόσπαση των εργαζόμενων, καθώς επίσης και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν μπορώ να κατανοήσω συντηρητικοί και φιλελεύθεροι να εγκρίνουν κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο κείμενο, γιατί στο κάτω τη γραφή καταστρατηγούν τις προσπάθειες των ίδιων του των εκπροσώπων μέσα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, δεν ήθελα να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση, λέει ο πρόεδρος Μάλκολμ Χάρμπορ, αλλά και ο Σουάμπ νομίζω ζήτησε πρώτο το λόγο. Όμως είναι ο Επίτροπος Μπαρνιέ εδώ και το απευθύνω το καλώς ορίσατε. Αν θέλετε να προβείτε σε συντομότατες δηλώσεις. Δεν έχω προετοιμάσει δήλωση, αλλά από την πλευρά της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Χριστιανών Δημοκρατών ε, να πω κάτι. Εμείς θεωρούμε ότι εξαντλητικός κατάλογος προσφέρει ασφάλεια δικαίου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να είναι το μενού του μεσημεριανού γεύματος προϋπόθεση για το αν θα σταλούν αποσπασμένοι εργαζόμενοι σε γειτονική χώρα. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης είμαστε ασφαλώς υπέρ της συνέχισης των ελέγχων στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλώς και πρέπει η υπόθεση Amazon στη Γερμανία να εξεταστεί σε βάθος. Τέτοια πράγματα δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν. Θέλετε να προσθέσετε πραγματικά κάτι σε αυτό. Κυρία Γκέπχαρτ, είναι απολύτως εσφαλμένο αυτό που λέτε. Οι τρει φιλελεύθεροι υποστηρίξαμε την τροπολογία της κυρία γέννη. Εσείς εδώ διαδίδετε εσφαλμένα μηνύματα και σα παρακαλώ να το παραλείψετε στο μέλλον. The will carry on. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και στην ΕΚΟΝ. Ελπίζω η συνάδελφος να εξακολουθήσει να εξετάζει αυτό το θέμα, παρότι κατανοώ την αποκοητευσή της. Έχουμε ζωντανό πολιτικό διάλογο στην την Επιτροπή μα. Πολλά διαφορετικά ζητήματα να εξετάσουμε και με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κ. Μισελ Είναι τακτικό επισκέπτη στην Επιτροπή μα. ήθελα να πω ότι η Επιτροπή μα μόλι ε, ψήφισε να δώσει εντολή ε, στου συζητητέ για την αμοιβή αναγνώριση προσόντων, ε, τη σύμβαση παραχωρήσεων και, τον, και τις οδηγίες τις οδηγίες για ε, τις δημόσιες προμήθειες. Για ε, τις διαπραγματεύσεις λοιπόν για όλα αυτά. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Δούμε στενά με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σημαντική εξέλιξη λοιπόν για την Ευρώπη και για την νομοθετική πράξη της ενιαίας αγοράς 1 και 2. Έχουμε μείνει λίγο πίσω βέβαια στα χρονοδιάγραμμα. Από την άλλη όμως η δουλειά μας ήταν ποιοτική και έτσι δεν λυπάμαι. Χαιρόμαστε που σας καλωσορίζουμε εδώ λοιπόν στο πλαίσιο ενός ε, δομημένου ε, διαλόγου για το πρόγραμμα εργασιών σας ε, για το υπόλοιπο της θητείας σας αλλά και για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτική μας θητείας. Ξέρω ότι πάντα ήσασταν ε, ιδιαίτερα συνεργάσιμος και πάντα μας δίνατε και μας ενημερώνατε για το πρόγραμμα εργασιών σας. Έχει ανοίξει ο κατάλογος ομιλητών. Ήδη πολλοί έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, όμως βεβαίως και σκιώδεις θα έχουν το λόγο και η κυρία Στάιλερ και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν μπορούν να το κάνουν. Επίτροπε Μπαγνιέ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Μάλκολμ, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που ξανασυναντιόμαστε εδώ σε αυτή την επιτροπή που για πολλούς λόγους είναι και η δική μου επιτροπή. Και να σας μιλήσω για τα όσα έχουμε κάνει και θα κάνουμε για να λειτουργήσει καλύτερα αυτή η μεγάλη ε, οικονομική, ανθρώπινη και κοινωνική κοινότητα που είναι η εσωτερική αγορά ακριβώς το πνεύμα που αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα και στα κείμενα που έχετε ενώπιόν σας. Για να μπω κατευθείαν στο ζήτημα των ε, προτάσεων που έχουμε υποβάλει στο πλαίσιο του Single Market Act 1 και 2, έχουμε και αυτά τα quick wins, όπως τα αποκαλώ, με τη μεταρρύθμιση των δημόσιων προμηθειών ε, και προτάσεων που έχετε αποφασίσει να υιοθετήσετε σε ό,τι αφορά τον τριμερή διάλογο τουλάχιστον. Συμμετέχετε με επαγγελματικό πνεύμα. Για τις δημόσιες προμήθειες αρχικά. Και η Αναβέλα έφυγε, αλλά την ευχαριστώ για τη δουλειά που έχει κάνει μαζί με τους υπόλοιπους ε, εισηγητές και συντονιστές. Η θέση μου είναι ότι οι εκάστοτε θέσεις μας δεν είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες κατά του τοπικού προστατευτισμού και, της, ε, και σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία δημοσίου-δημοσίου. Εδώ λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο για να απλουστεύσουμε αυτές τις διοικητικές συμβάσεις που είναι ιδιαίτερα επαχθείς ε, ε, σε βάρος ε, των επιχειρήσεων, να ενισχύσουμε την ευστερική αγορά και για να καταστούν αυτές οι δημόσιες προμήθειες πιο καινοτόμες, χωρίς αποκλεισμούς και προστατεύοντας το περιβάλλον. Σε ό,τι φορά τις συμβάσεις παραχώρησης, και εδώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή Φιλίπ Ζουβά και τους συντονιστές. Γνωρίζετε γιατί παρουσίασα και επέβαλα αυτό το κείμενο ταυτόχρονα με τις δημόσιες προμήθειες, γιατί δεν υπήρχε ένα ελάχιστο κανονιστικό πλαίσιο για, για αυτό το είδος ε, συμβάσεων, όπως είναι οι συμβάσεις παραχωρήσεων, που ε, χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο. Και χρειαζόμασταν ένα τέτοιο ελάχιστο κανονιστικό πλαίσιο για να υπάρχει διαφάνεια και για να μην υπάρχουν διακρίσεις στην ενιαία αγορά, αλλά και για την προστασία των ε, πολιτών. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, για τη δουλειά που έχετε κάνει. Πολύ συχνά έχω αναφερθεί στην ε, σημασία των δημοσίων διαβουλεύσεων, των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου εδώ στο Κοινοβούλιο είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα λοιπόν αυτός ο δημόσιος διάλογο και τα ζητήματα που τίθενται εκεί. Πολλές φορές υπάρχουν και λανθασμένες ε, κατηγορίες και θα είμαι εξαιρετικά σαφή εδώ. Δημοσίω ενώπιόν σας, εκ μέρους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ως πολιτικός και πολίτης, Κυρίε και κύριοι, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει καμία ιδιωτικοποίηση του ύδατο ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον. Και αυτή η οδηγία δεν έχει τέτοιο στόχο, ούτε τέτοιες επιπτώσεις θα έχει αυτή την ε, υποχρεωτική ιδιωτικοποίηση των ε, υπηρεσιών ε, πόσμου ύδατος, ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον επαναλαμβάνω. Δεν θα μπορούσα να σας ε, υποβάλω ένα τέτοιο κείμενο. Αντιθέτως, στο κείμενο όσο έχει, αναγνωρίζουμε ξεκάθαρα την ελευθερία των κρατών μελών και επανεπιβεβαιώνουμε την αυτονομία των τοπικών αρχών σε αυτόν τον τομέα. Οι τοπικές αρχές είναι αυτές που καθορίζουν ποιες είναι οι υπηρεσίες κοινή ωφελία και επιλέγουν ελεύθερα τον καλύτερο τρόπο διαχείρισής τους. Αυτό διασφαλίζεται από τη συνθήκη, το πρωτόκολλο 26 και κανένας ευρωπαϊκός νόμος δεν μπορεί να ε, αντιβαίνει σε μια τέτοια θεμελιώδη αρχή. Και σας λέω εδώ κυρίες και κύριοι και πάλι ε, επανεπιβεβαιώνω την βούλησή μου και τη δέσμευσή μου να τηρηθεί αυτή η αρχή. Είχα την ευκαιρία να το συζητήσω με πολλούς εξημών και με τον κύριο Σβόμπ. Ε, αναγνωρίζω και γνωρίζω μάλλον αυτές τις πρωτοβουλίες των πολιτών με τις υπογραφές, τη συλλογή υπογραφών και θεωρώ πολύ καλές αυτές τις ε, και μπορώ να σα πω μάλιστα ότι εγώ είμαι έτοιμος να υπογράψω αυτή την ε, αίτηση. Κανένα πρόβλημα που θα διασφαλίζει δηλαδή τον δημόσιο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και την ποιότητα του ύδατο. Σε ένα σημείο μόνο διαφωνώ με αυτή την αίτηση. να βγουν υπηρεσίε ύδατο από του κανόνε ε, τη εσωτερική αγορά. Αυτό δεν θα αποβεί σε όφελο ούτε των καταναλωτών, ούτε των πολιτών, ούτε των φορολογουμένων. Όταν δηλαδή οι συμβάσει ε, ε, γίνονται, ε, συνάπτονται με τις τοπικές αρχές, θα πρέπει αυτό να γίνεται με διαφάνεια, να υπάρχουν ευρωπαϊκά κριτήρια σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ύδατο, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδάλλως ένας ε, Φιλανδό, Γερμανός ή Γάλλος επίοικο που πάει σε μια άλλη χώρα δεν ε, ε, έχει εξασφαλισμένη ποιότητα ύδατο. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κοινοί κανόνε. Μόνο αυτή την επιφύλαξη λοιπόν έχω. Εκτός από αυτό το σημείο τα υπόλοιπα τα προσυπογράφω. Βεβαίως το νερό να διασφαλίζεται ότι θα είναι δημόσιο αγαθό. Ε, ρητέ πεπιθήσεις λοιπόν ε, ως προς αυτά τα σημεία. Υπάρχουν βεβαίως κάποια ερωτήματα ή ενδεχομένως ε, παρανοήσεις. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να διασκεδάσω τις ανησυχίες που εκφράζονται στην Αυστρία, στη Σλοβενία, στη Γερμανία για αυτό το θέμα. Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, είμαι διατεθειμένος να στηρίξω κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων που θα ξεκινήσουν, να υποστηρίξω λοιπόν νέες διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο. Ε, συνομίλησα και με τον εισηγητή κύριο Ζουβάν που έκανε κάποιες ε, προτάσεις και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις συζητήσεις που έχω κάνει με τον κύριο Σουά πολλές φορές, με την κυρία Γκεμπάρτ ή την κυρία Ρούλε. Ποια είναι η κύρια δυσκολία. Στη Γερμανία έχουμε το λεγόμενο Stadtwerke, με πολλές δραστηριότητε, πολλούς ε, κλάδους. Αυτές οι επιχειρήσεις ως παραδοσιακή πάροχοι έχουν ένα προστατευόμενο ε, δημόσιο μονοπόλιο κατά την ε, διανομή του ύδατος στις κοινότητες. Με μία ή άλλη μορφή αυτό υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πρόκειται να θέσουμε να αμφιβόλο αυτό το καθεστώς. Ποτέ. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Ταυτόχρονα Πολλέ φορές αυτές οι επιχειρήσεις ε, δραστηριοποιούνται σε τομείς που είναι ανοιχτοί ε, στον ανταγωνισμό, στην ενέργεια, στις μεταφορές. Εκεί μιλάμε για δημοτικές ε, τέτοιε επιχειρήσεις, τα και που έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα. Και ο κανόνας που δεν τον εφήβρα εγώ, αλλά είναι το δικαστήριο του Λουξεμβούργου και με βάση και με την νομολογία τη γερμανική, με απόφαση του ε, δικαστηρίου του Αμβούργου, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι αυτές οι επιχειρήσεις, ακόμα και με ιδιωτικά κεφάλαια, μπορούν να υποφελούνται άμεσων συμβάσεων χωρίς ε, ανταγωνισμό και χωρίς διαφάνεια εκ μέρους των ε, Δήμων. Υπό δύο προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή, όταν πράγματι ελέγχονται από το Δήμο και όταν το 80% των δραστηριοτήτων τους αποβαίνουν προς όφελος του Δήμου. Κατάλαβα όμως το πρόβλημα ακούγοντάς σας και ακούγοντας και τους εκπροσώπους των γερμανικών και αυστριακών δήμων είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι πολυκλαδικές, μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς που είναι ανοιχτοί ε, στον ανταγωνισμό και σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές δεν πληρούν το κριτήριο το 80%. Και έτσι χάνουν αυτό το καθεστώς. Θέλω λοιπόν να βρω μια δίκαιη και εξισορροπημένη λύση μαζί σα για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα και για να μην υπάρχουν βεβαίω στρεβλώσει του ανταγωνισμού. Γι' αυτό και συνομίλησα με τον ε, εισηγητή κ. Ζουβά που μου πρότισε, πρότεινε μια νέα διατύπωση. Ο κανόνας του 80% λοιπόν να ε, ισχύει μόνο στις... Ε, μόνο σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε που συνδέονται με το νερό και όχι στις συνολικέ δραστηριότητε. Μόνο λοιπόν στις δραστηριότητε που συνδέονται με το νερό για το Δήμο. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση πρέπει να έχει μια διαφορετική διαχωρισμό, ένα διαρθρωτικό διαχωρισμό ή μια διαφορετική εταιρική ευθύνη ενώπιον του Δήμου. Έτσι λοιπόν μπορούμε να τροποποιήσουμε τον ορισμό των λεγόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων ε, για τους ε, γειτονικούς ε, όμορους δήμους, για παράδειγμα, γιατί πολλές φορές αυτοί οι δήμοι συνεργάζονται με τους όμορους δήμους. Και ίσως πρέπει να το εξετάσουμε από την πλευρά μιας γεωγραφικής συνοχής. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές που θα μπορούσα να στηρίξω. Έχοντας ε, έρθει σε επαφή με τον εισηγητή και με άλλους συναδέλφους. Αυτό το κείμενο λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσει ξεκάθαρα ότι ε, οι Δήμοι μπορούν, έχουν την ελευθερία να παράσχουν οι ίδιοι το, ε, Υπηρεσίε νερού προς τους ε, δημότε τους, είτε να αναθέτουν αυτές τις υπηρεσίε σε κάποια άλλη επιχείρηση. Αλλά βεβαίω, αν ε, παραχωρηθεί σε μια άλλη ε, επιχείρηση, τότε θα πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια της διαφάνειας και των μη διακρίσεων. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, και εδώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό διαφάνειας των κλειστών επαγγελμάτων ή σε ό,τι όπου υπάρχουν ε, σημαντικές εξελίξεις. Θεωρούμε ότι ο διάλογος που θα ξεκινήσει τριμερός θα είναι επικοδηματικός. Ε, για ορισμένα κλειστά επαγγελμάτα πρέπει να βρεθούν συμβαστικές λύσεις, όπως είναι συμβολιογράφοι, όπου οι απόψεις ε, διείστανται και στο Συμβούλιο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε οριστική απόφαση. Σε αυτό το σημείο όμως θα διατηρήσουμε επικοδηματική στάση ως Επιτροπή. Οι εκτινίατροι, οι ΜΕΕΣ και γνωρίζω την ε, καθημερινή ε, πραγματικότητα αυτών των εξαιρετικά δύσκολων επαγγελμάτων. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια λύση Έχουν ε, εκφραστεί αντίθετες απόψεις ως προς ε, αυτές τις προτάσεις λοιπόν και πρέπει να επικεντρωθούμε και στις ε, θεμελιώδεις απαιτήσεις που συνδέονται με αυτά τα επαγγέλματα και να δούμε και κάποιες στοιχές της κατεξοδότησης πράξης. Τέλος, σε ό,τι αφορά την κινητικότητα της οδηγίας, που αναφέρεται στην οδηγία, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κανόνας και ίσως θα πρέπει να επανεξετάσουμε στο μέλλον αυτή την πτυχή, ε, κρατώντας πάντα υπόψη την ε, απλότητα της διαδικασίας αυτής της ε, κινητικότητας. Για να επιστρέψουμε και στο σημείο των 5 ετών, ε, υπάρχει ένας προβληματισμός σε αυτό το σημείο και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με το Συμβούλιο για να εξεύρουμε μια εξισορροπημένη λύση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, αυτά τα δύο μεγάλα θέματα των δημοσίων προμηθειών και των ε, επαγγελματικών προσόντων. Θα πρέπει να αφαιρθώ και γενικότερα ε, στο χάρτη πορείας του SMA 1 και 2. Για το SMA 1, το Single Market Act, έχουμε την εφαρμογή όλων αυτών των βασικών δραστηριοτήτων, 12 τον αριθμό Δύο από αυτέ έχουν υιοθετηθεί επισήμω από το Κοινοβούλιο. Τρεις ακόμα ε, αποτελούν αντικείμενο πολιτικής συμφωνίας και θα υιοθετηθούν επισήμω ε, τις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της Ιρλανδική Προεδρίας να, ε, να κλείσει το θέμα της οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφέ και για τους ε, λογιστέ. Και μετά, 12 από τις 12 δραστηριότητες του ε, SMA1, σε αυτές αναφέρομαι, αλλά δεν αναφέρομαι στις 50 επιπλέον ε, πρωτοβουλίες ε, του SMA1 που θα ήταν καλό να προχωρήσουν. Ένα πολύ σημαντικό είναι η οδηγία περί Εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι, να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που έχουμε Έχουμε και την ανακοίνωση πλαίσιο του προηγούμενου Ιουνίου, βάσει της οποίας χρειαζόμαστε ε, έντονη κινητικότητα και κινητοποίηση μάλλον σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές χώρες. Το επανέλαβα και προχθές. Και χαίρομαι και για την ε, προσοχή που δίνετε σε αυτό το τομέα στην Επιτροπή σας. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Άκουσα και πολύ καλά λόγια για την ακρόαση που ε, χθε. Έχουμε και περαιτέρω δραστηριότητε, ομάδα υψηλού επίπεδου για ε, αυτό το θέμα. Η πρώτη συνεδρίαση θα λάβει χώρα ε, στις αρχές Μαρτίου. Δεύτερη δραστηριότητα 31 Ιανουαρίου ε, υιοθετήθηκε από τους Επιτρόπους. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το ε, ελληνικό εμπόριο. Και μετά η πράσινη βίβλος ε, για τις ε, παράνομες εμπορικές πρακτικές. Και θα ήθελα η Επιτροπή σας να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά το SMA2 και πάλι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση, παρότι ίσως καθυστερούμε, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες προτάσεις μέχρι το φθινόπωρο για να έχετε και εσείς το χρόνο μέχρι την επόμενη άνοιξη να προχωρήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο προς την υιοθέτηση των 12 νέων προτάσεων του SMA2. Τρεις προτάσεις έχουν, ακόμα, έχουν ήδη τεθεί επιτάπητος σε ό,τι αφορά την αφαιρεγγιότητα, τρίτο πακέτο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και την προηγούμενη εβδομάδα το ε, πακέτο για τη γενική ασφάλεια ε, προϊόντων και της εποπτείας της αγοράς. Έχουμε ε, ένα σχέδιο δράσης για το Eures, τη θύρα Eures και για το τρίτο πακέτο της ενέργειας. Και τέλος, επιβεβαιώνω και πάλι τη δέσμευσή μας στο πλαίσιο του SMA2 να σας παρουσιάσουμε μια πολύ σημαντική για μένα ε, πρόταση, δηλαδή τη διαφάνεια των ε, τραπεζικών τελών, την τραπεζική κινητικότητα και σε ό,τι αφορά την ε, σε φορά του, του διαδικτύου υψηλή ταχύτητα. Είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό για μένα στο πλαίσιο τη εμόρφωση της ψηφιακής μα αγορά. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε ό,τι αφορά την ε, αγορά και πώληση στο διαδίκτυο. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον Παύλο Αριάς και Σεβάρια για τις εργασίες ε, που έχουν καταβάλει για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Επιτροπή σας. Η Επιτροπή έχει θέσει έναν ορίζοντα μέχρι το 2015 για τις ηλεκτρονικές ε, πωλήσει. Εδώ και ορισμένου μήνες έχουμε παρουσιάσει ε, τις πρωτοβουλίες μας για την παράδοση των ε, δεμάτων και τον επόμενο μήνα θα παρουσιάσω έκθεση για την πρόοδο των εργασιών μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ενιαία ψηφιακή αγορά, έχουν τεθεί επιτάπητος πολλές προτάσεις, συλλογικές συμβάσεις, πνευματικά δικαιώματα, License in Europe και άλλες προτάσεις πρόκειται να έρθουν για την ε, ε, ηλεκτρονική τιμολόγηση ή τις ε, υπηρεσίες πληρωμών. Ευρύ φάσμα λοιπόν, αλλά θέλω να σας δώσω αυτή την ιδέα της έννοιας και ο πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε σε αυτό προηγουμένως, ότι υπάρχει το βασικό περιεχόμενο του SMA 3, στο οποίο θα ήθελα να εργαστώ μαζί σας. Εάν σήμερα το... Ε, αν φέτος το φθινόπωρο διαμορφώσουμε ένα Single Market Act 3, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις προτάσεις των συναδέλφων, θα πρέπει όπως και να έχει να έχουμε προχωρήσει με την, στην υλοποίηση του Single Market Act 1 και 2. Γιατί όταν όλες οι προτάσεις ε, γίνονται στον αέρα, τότε δεν είμαστε και αξιόπιστοι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό για το 2013. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ ε, στον δημόσιο διάλογο και στη διακυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα για τη διακυβέρνηση, να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Σουάμπ για την έκθεσή του, για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του scoreboard σε ό,τι αφορά την ε, ενιαία αγορά στο διαδίκτυο, που θα δημοσιεύσουμε το καλοκαίρι. Συμφωνώ με την ιδέα μια συνδιάσκεψη που θα αφορά ακριβώ το ζήτημα τη διακυβέρνηση, ε, που θα συνδιοργανωθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενδεχομένω ε, την ε, επερχόμενη Λιθουανική Προεδρία το Σεπτέμβριο. Για να υπάρχει αυτό το peer pressure μεταξύ των κρατών μελών, την προηγούμενη Τρίτη παρουσίασαμε το τελευταίο scoreboard ε, σε ό,τι αφορά την συμμόρφωση με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ε, και βλέπουμε ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στους τελευταίους μήνες με νέα ε, μείωση σε ό,τι αφορά το έλλειμμα μεταφοράς που, νομοθεσία, της νομοθεσίας που είναι πλέον στο 0,6% σε σχέση με 1,2% που ήταν πέρσι. Και πάλι σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την ε, συμμετοχή της ε, σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση νομοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά που θα ολοκληρωθεί τον επόμενο Σεπτέμβριο. Και βεβαίως να υπενθυμίσω και τα όσα θα διοργανώσουμε στην Κρακοβία. Την εβδομάδα της εσωτερικής, της ενιαίας αγοράς, όπου θα κάνουμε τον απολογισμό ε, της ενιαίας αγοράς. Θα έχουμε ένα μήνα λοιπόν για να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό του Single Market Act 1. Τέσσερις εβδομάδες λοιπόν ε, από 20 Σεπτέμβρη με 20 Οκτώβρη. Τέσσερις εβδομάδες θα έχουμε στη διάθεσή μας να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό ε, μεταξύ μικρών ομάδων, θεματικών ομάδων ε, που θα εκπροσωπούν όλα τα κρατημέλη, θα βρεθούν εδώ στις Βρυξέλλες για τους πολίτες και τις τράπεζές τους, ε, την ε, ε, ψηφιακή αγορά. Πολλά πολλά είναι τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια αυτών των 4 εβδομάδων. Τρία κείμενα θα σας υποβάλω. Πρώτα ο πίνακας για το Single Market Act 1 και 2, το πρόγραμμα εργασιών μας για το 2013 που αφορά συγκεκριμένα την Επιτροπή σας και τέλος ε, το scoreboard, scoreboard 26 για την ενιαία αγορά που αναφέρεται στο, στα ποσοστά μεταφοράς νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Well, it's clear that you're going to keep us... Κύριε Επίτροπε, ήταν ξεκάθαρο ότι θα είμαστε αρκετά, θα έχουμε αρκετά περιμένει ατζέντα σύμφωνα με όσα μας ε, ανακοινώσατε. Χαιρόμεθα ιδιαίτερα για πολλά από όσα μας είπατε και ιδίως αυτή την ιδέα που αναφέρατε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για την ενιαία αγορά και ιδιαίτερα στα πλαίσια της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, κάτι που ζήσαμε και εμείς. Βάλτε λοιπόν στην ατζέντα σας όλοι αυτή την ημερομηνία για τη διάσκεψη για την ιστορική αγορά πριν τι εκλογέ. Πολύ σημαντικές Οι επίσης επίση ζητούν αυτό το θέμα και θα πρέπει να δουλέψουμε με πρωτοβουλίες. πρωτοβουλίε. Ε, δεν έχουμε εκθέσει αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε πάρα πολύ υλικό. Μα δώσετε πολύ σημαντικό υλικό ενώ σε αυτές τις Συνάδελφοι, η κομισ... ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή δεν μπορεί να μείνει πολύ περισσότερο μετά τι 11 και 14, αλλά Ξέρω ότι έχουμε 15 συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Που κα... Αν ακόμα και σας το λόγο για ένα λεπτό, σίγουρα θα καλύψετε αυτό το χρόνο που μας μένει. Να δώσω κατευθείαν τον λόγο στους συντονιστές ή ε, οπωσδήποτε απαραίτητο να δώσω τον λόγο κατευθείαν στους συναδέλφους. Λοιπόν, όσοι δήλωσαν το διάθεση να μιλήσουν πρώτοι, σε αυτούς θα δώσω το λόγο. Και ανάλογα με το πόσο λακωνική θα είστε, πιο πολύ θα πάρω το λόγο. Η κυρία Στάιλερ. Ρόσφορ. Κυρία Ελεγκρίπ, αυτός είναι ο πρώτος γύρος. Ας πάρουμε τέσσερις ομιλητές. Και Σαλαμάγιο. Αυτή είναι οι τέσσερις πρώτοι αγορητές. Παρακαλώ λοιπόν να είσαστε έτοιμοι να πατήσετε το κουμπάκι τη της Λοιπόν, κύριε Σάλλον, πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία του Επιτρόπου. φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα τη αδειοδότηση και το copyright. Είχαμε μια συνέντευξη πριν από κάποιε εβδομάδε για αυτό το θέμα και ιδιαίτερα το θέμα τη πρόσβαση των βιβλιοθηκών σε βιβλία με ηλεκτρονική μορφή. Δεν θέλουμε ένα ηλεκτρονικό apartheid για τι βιβλιοθήκε. Αυτή τη στιγμή πολλοί εκδότε δεν επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες να έχουν πρόσβαση στην ε, ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων. Πιστεύω ότι είναι καλό σε έξι μήνε να μα ενημερώσετε και πάλι για αυτό το ζήτημα και καλό να κάνετε κάτι στην κοινή σα διεύθυνση αυτού. Uh, καλό παράδειγμα, ο κύριο Ρόσφορντ. Ευχαριστώ και εσά και Επίτροπε. Όλοι αναγνωρίζουμε τις πρόοδους της ενιαίας αγοράς. Καμιά φορά, ωστόσο, ορισμένα ενοχλητικά αμαυρώνουν την εικόνα. Όπως αυτό το ατυχές γεγονός της ανάμιξης κρέατος ε, αλόγου σε βόλιο, που εν τέλει δείχνει ότι εκεί όπου ανακατεύονται πολλές χώρες τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί ανοίγουν τον δρόμο στην κερδοσκοπία. Δεν είναι πρόβλημα προστασίας της υγείας, αλλά της αληθείας των ισχυρισμών επί της ετικέτας. Είμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Είναι απαραίτητο η επικοινωνία σχετικά με την ενιαία αγορά να ξαναβρει μια σωστή ισορροπία υπέρ του καταναλωτού. Και στα έγγραφα που μας ε, δίνεται σήμερα στοχεύουν ιδιαίτερα στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις που θεωρώ πράγματι είναι πολύ σημαντικές, αλλά δεν αρκεί. Και η εικόνα που δόθηκε στην ακρόαση για τις υπηρεσίες για τις οποίες μιλήσατε προηγουμένω ήταν καθαρή. Σήμερα οι καταναλωτές δεν βλέπουν ακόμα καθαρά με ποιον τρόπο θα αρθούν τα εμπόδια. Με ποιον τρόπο να μπορεί να αγοράζει σε άλλη χώρα από τη δική του, του επιτρέπει να εποφελείται από ανταγωνιστικές τιμές. Μέχρι από εδώ, από εδώ και μέσα στον επόμενο χρόνο πρέπει να μας δώσετε πυρομαχικά για να μπορέσουμε να αποδείξουμε στους καταναλωτές ότι κάτι κάνουμε. Μην κάνετε σχόλια να κάνετε ερωτήσει. Αν ναι, στην τελευταία σα φράση είχατε ένα, ένα έμεσο ερώτημα. Και εν πάση περιπτώσει είχατε πει και άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση με την Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά το σχόλιο ήταν καλό. Κύριε κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τι εισαγωγικέ σα παρατηρήσει, Δύο ερωτήσει. Πρώτον, επικοινωνία για την ενιαία αγορά προς τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας. Σημαντικό διακύβευμα Σημαντικέ οι πρόοδοι τη ενιαία αγορά, ωστόσο και οι πολίτε, όχι μόνο οι επαγγελματίε και επιχειρήσει, αλλά και οι καταναλωτέ εν τέλει πρέπει να είναι ενήμεροι για να γνωρίζουν ποια είναι τα κεκτημένα, τα διακυβεύματα και τα δικαιώματά του, για την κινητικότητα, για ε, επαγγελματικά προσόντα, αναγνώριση κτλ. Όλα αυτά πρέπει επιτέλου να φτάσουν μέχρι τον καταναλωτή. Τι γίνεται τώρα με, το, με την πύλη Europe, το πόρταλ αυτό. Είναι ικανοποιητική η λειτουργία της. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς. Δεύτερο, Κίνα και, τις, και την πρόσβασή της στις δημόσιες προμήθειες. Και το αντίθετο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινέζικη αγορά, κυρίως για υλικό τηλεπικοινωνιών, που γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση των επιχειρήσεων μας στην κινέζικη αγορά. Ευχαριστώ, Σάλντε Μόζερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αλλά και εσάς κύριε Επίτροπε. Δύο σχόλια. Αφενός χαίρομαι που θα γεννούν συστάσεις για πιο υπεύθυνη διαφήμιση στο διαδίκτυο καθώς επίσης και για, ιδίως για τα τυχερά παιχνίδια. Στην Δανία βλέπω για παράδειγμα ιδιαίτερα επιθετική διαφήμιση για τα τυχερά παιχνίδια. Και σωστό είναι αυτά τα πράγματα να ρυθμιστούν, μου φαίνεται καλό. Δεύτερο, ψηφιακή αγορά. Σωστό. Αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου. Χρειαζόμαστε ωστόσο και μια πρωτοβουλία για να είναι πιο καθαρές και οι ε, ενδείξεις για τις κεραίες στα κινητά μας τηλέφωνα υψηλής ευφύειας. Um, Μάλιστα, να δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει, αλλά σημειώνω και εγώ γιατί δεν θα καταφέρω να δώσω το λόγο σε όλους. Ο κ. Βονίου και ο κ. Ζουβά να πα τις επόμενες ερωτήσεις όσες ηγητές. Κύριε Κορέτσα Μπίλτ, λόγω της Εχθέ Ο κύριο Άρια επίσης να πατήσει για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτοί είναι τέσσερι σημαντικοί αγορητέ συναφεί με το θέμα. Και μετά θα δούμε με του συντονιστέ και του λοιπού. μετά τι απαντήσει του Επιτρόπου. Απλά σα λέω να είστε έτοιμοι για το ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και να τηρήσω την ε, ίδια πειθαρχία που απαιτεί ο πρόεδρος από εσάς. Η κυρία Στάιλερ ανέφερε ε, τα δικαιώματα δυνατικής ιδιοκτησίας. Βεβαίως εδώ έχουμε ορίσει μια στρατηγική που σας έχει προτείνει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σύγχρονη προστασία, ούτως ώστε να ευθυγραμμιζόμαστε και με τις σημερινές συνθήκες. Η σημερινή εποχή είναι η εποχή του διαδικτύου. Ήδη έχουμε εφαρμόσει τμήματα της στρατηγικής για τα ορφανά έργα, ας πούμε, είναι τμήμα της ε, πρότασης ε, για την ε, ψηφιοποιημένη πρόσβαση. Αυτό έχει ήδη υιοθετηθεί και έχει τεθεί σε ισχύ. Η συλλογική διαχείριση ακόμα συζητείται με αυτό που ανέφερα για την πολυεδαφική άδεια. Και για να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα, σε ό,τι αφορά με την κυρία Κρόσα αυτά που ανέφερε, εμείς έχουμε ξεκινήσει ένα συμβατικό έργο ε, με ένα πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένα ζητήματα που μπορούμε να, όπου μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο μέσω αυτών των συμβάσεων και αυτό έχει ξεκινήσει ως εγχείρημα τις τελευταίες ημέρες. για παράδειγμα, ένας ε, πολίτης ε, που περνά τα σύνορα έχει μία ε, συνδρομή στη χώρα του να μπορεί να τη χρησιμοποιεί και στη γειτονική χώρα, κάτι που το οποίο δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να επιτύχουμε με το λεγόμενο Licensing Europe. Ο κ. Ροσφόρ ανέφερε την κρίση της επιστηστικής ασφάλειας που παρατήρησαμε σε πολλές χώρες. Πρόκειται ε, για μια απάτη ουσιαστικά. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ποιος ήταν υπεύθυνο για αυτή την απάτη. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες ε, στους υπευθύνους. Εμείς επαναπροσανατολίζουμε τη δράση μας όταν δεν είναι επαρκής προς τους καταναλωτές ε, και ο συνάδελφος Μπόρκ είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε όλα αυτά. Έχει ε, εντοπίσει και συγκεκριμένα εργαλεία για την προστασία των καταναλωτών. Εμείς έχουμε εξαιρετικά επικοδομητικές ε, σχέσεις με τον Επιτρόπο Μπόρκ για αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές υποβάλλω τέτοιες προτάσεις και κύριε Ροσφόρ, επιβεβαιώνω ότι πέραν των όσων έχω κάνει ε, σχετικά με πολλές ε, οδηγίες περί χρηματοοικονομικών για την προστασία των ε, καταναλωτών, ε, ένα επίπεδο προστασίας που δεν το είχαμε σε τα τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα, ε, σύντομα θα κάνουμε μια πρόταση που αφορά τη διαφάνεια των τραπεζικών τελών, που αφορά εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, και σε ό,τι αφορά την τραπεζική κινητικότητα. Επίσης, για το επιστημιστικό ζήτημα, βεβαίως και μπορούμε να πάμε παραπέρα. Για να πάμε πέρα από την ίχνη λασιμότητα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προπαρασκευασμένα ε, τρόφιμα, πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται. Οι καταναλωτές ε, δικαιούνται να γνωρίζουν και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Δεν πρέπει να υπάρχει ο φόβος αυτής της διαφάνειας. Η κυρία Λεγκρίπ αναφέρθηκε και εκείνη στους ε, πολίτες, όπως έκανε και ο κύριος Ροσφόχ. Ε, η πύλη New Europe ε, που αναφέρατε, σε ό,τι αφορά την πρακτική υπεράσπιση των δικαιωμάτων πολιτών και επιχειρήσεων που σε αυτή την επίλη μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται και να προσανατολιστούν προς ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως είναι η ενιαία θηρίδα ή το Solvit, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ε, ανέφερα στους υπουργούς ε, την αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων ε, που θα ενισχύσει την εγκύτητα των ευρωπαϊκών θεσμών και των Βρυξελών Προ του πολίτες. Θα νιώθουν πολύ πιο κοντά οι πολίτες με του Ευρωπαϊκού θεσμού χάρη σε αυτά τα εργαλεία. Ήδη υπάρχουν τέτοια μέσα που επιτρέπουν... Ε, υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου ε, υπάρχει πολύ στενή συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών διαφορετικών κρατών μελών, επιχειρήσεων που έχουν ένα αίτημα να κάνουν σε σχέση με τις αρχές άλλων χωρών το λεγόμενο IMI. Ε, αυτό λοιπόν ε, βοηθά πολύ τους πολίτες. Έχουμε 15.000 ε, χρήστες κάθε μέρα στο αυτό το U-Europe και ο αριθμός τους αυξάνεται καθημερινά. και με την πολύ καλή ορατότητα που έχουμε διασφαλίσει, με την χρήση για αξιοποίηση των συστημάτων δικτύωσης. Αναφερθήκατε στην Κίνα η Κίνα δεν ε, συμμετέχει στο GPA, Government Procurement Agreement, ε, που συνήθει στα τέλη του, της προηγούμενης χρονιάς και προτιμούμε, προσπαθούμε να πείσουμε τους εταίρους μας που συμμετέχουν στο GPA να ανοίξουν περισσότερο τις ε, αγορές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, κυρία Λογρήψ, σας Υπενθυμίζω ότι έχουμε παρουσιάσει ένα μέσο για την αμοιβαιότητα των δημοσίων προμηθειών. Νομίζω ότι είχατε και τον αρμόδιο επίτροπο για αυτά τα ζητήματα. Όχι για να κλείσουμε μόνο τις, ε, τις αγορές μας, όχι για να κλείσουμε μόνο τις αγορές μας, για να ανοίξουν και οι αγορές των άλλων, να είναι αμοιβαίο αυτό το άνοιγμα. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα ε, κλείσιμο, αν θέλετε, ένας αποκλεισμό ορισμένων ε, τομέων στην Ευρώπη, όπως συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ, ας πούμε, αλλά να γίνει με συντονισμένο και ομογενή τρόπο. Αυτό το GPA λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο συντονισμένο και συνεκτικό στην Ευρώπη. Και με την Κίνα συνεργαζόμαστε προκειμένου να προσχωρήσει στην συμφωνία αυτή. Κυρία Σαλντομεζέ αναφέρθηκε στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο που παρουσιάστηκε, παρουσιάσαμε στις 23 Οκτωβρίου του 2012 το πρόγραμμα, το σχέδιο δράσης μας για τη τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Χθε νομίζω εδώ με τον κύριο Φόξ αναφέρθηκαν πέντε βασικές προτεραιότητες. Ε, το, τα, τα εθνικά ε, προγράμματα και σχέδια δράσης, η βελτίωση των, ε, των επαφών, ε, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εθνικών αρχών, η προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα των νέων, που είναι και οι πιο ευάλωτοι απέναντι σε αυτά τα δίκτυα, η πρόληψη της απάτης και του ξεπλήματος χρήματος και κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η διασφάλιση της ακαιρεότητας του αθλητισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινός πυρήνας ε, για την καταπολέμηση ε, τέτοιων φαινομένων όπως είναι το στήσιμο παιχνιδιών, αλλά και για να καταπολεμήσουμε και τον εθισμό, να προστατεύσουμε τους ανηλίκους. Σίγουρα, σε ό,τι αφορά αυτή την ταχύτητα πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις. Και θα συνεργαστούμε και την κυρία Κρούς για να εξετάσει ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Okay, that's a big variety of questions πολλές και ποικίλε ερωτήσεις. Ήδη καλύψαμε πολλά θέματα, οπότε θα περάσουμε σε ένα επόμενο γύρο παρεμβάσεων ενό λεπτού που θα είναι οι εισηγητές σύν ο πρόεδρος μας Αυτό είναι το κριτήριο επιλογή Κ. Βανιού, Ζουβάου, Κοράτσα Πίλτα και Αρία Για ένα λεπτό. Κυρία Βανιού. Ε, θα προσπαθήσω να τα πω πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Απαντήσατε ήδη σε τρεις ερωτήσεις που επιθυμούσα να θέσω. Ξεχάστε Είπατε για την οδηγία επαγγελματικών προσόντων, για ορισμένους επαγγελματικούς τομείς. Αυτό θα χρειαστεί και άλλη συζήτηση. Ένα πρόβλημα που έχω μετά τις ψηφοφορίες είναι το πρόβλημα των επαγγελματικών ασφαλίσεων σε περίπτωση κινητικότητας των επαγγελματιών. Είναι και αυτό θεμελιώδου σημασίας για να δώσουμε και να προσφέρουμε και εμπιστοσύνη δηλαδή στους ίδιους τους επαγγελματίες για την ασφάλεια δικαίου αλλά και στους πολίτες έτσι ώστε να έχουν καλύτερες πληροφορίες των όσων ποιούνται χρήση των επαγγελμάτων αυτών. Και απευθύνομαι σε εσά την Κομισιόν διότι το πρόβλημα των ασφαλίσεων είναι πολύ σημαντικό και για την ώρα υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν από μια χώρα σε άλλη γιατροί για παράδειγμα, καλούνται να ασφαλιστούν δύο φορές, κάτι το οποίο δεν είναι καλό ούτε για τους ίδιους ούτε για τους πολίτες. Και με συγχωρείτε, ξεπεράσατε το λεπτό σας. Ε, ο κύριος Ζουβά. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, μόλις μιλήσατε για την αναφορά που υπο, βρίσκεται στη φάση της υπογραφής τώρα για τις ε, συμβάσει παραχωρήσεων, ε, στι υπογραφή σε διάφορε χώρε μέλη. Υπάρχει όντω κίνδυνος ιδιωτικοποίησεω της παροχής πόσιμου ύδατος. Εσεί κάνετε ορισμένε προτάσει, θα επανέλθω σε αυτέ, και υπάρχουν και μια κατηγορία ανθρώπων που χρησιμοποιούν την συλλογή αυτή υπογραφών για πολιτικού στόχου. Στη Γαλλία λέμε, άμα θέλει να ξεφορτωθεί το σκύλο σου, πε ότι έχει λύσα άμα θες να ξεφορτωθεί στην Ευρώπη, πες ότι πάει κάτι να ιδιωτικοποιήσει. Είναι περίπου το ίδιο. Αφενός λοιπόν να καθησυχάσουμε αυτούς που φοβούνται την ιδιωτικοποίηση, δεν νομίζετε ότι μπορούμε επισήμω να πούμε μέσα στο ίδιο το κείμενο του νομοθετήματος για να έχει και κάποια νομική βαρύτητα, να πούμε ότι αυτή η οδηγία περί παραχωρήσεων δεν θα οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση. Να είναι λοιπόν στο άρθρο πρώτο, να, είναι, να έχει βαρύτητα νόμου. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την οδηγία υπηρεσιών. Ευχαριστώ που μνημονεύσατε τη χθεσινή ακρόαση που ήταν πράγματι πολύ ωραία. Όλοι θα σας υποστηρίξουμε στην πρότασή σας για μηδενική ανοχή για τη μη σωστή εφαρμογή. Ερώτηση, τι μπορεί να κάνει κανείς με την έκθεση του Κοινοβουλίου ώστε να σας βοηθήσουμε να συνεργαστούμε με τρόπο επικοδομητικό ώστε να αποδώσουμε ξεκάθαρα αποτελέσματα πίεσης επί των χρόνων μελών. Έχουμε την έκθεση ΣΟΑΜ για την ε, διακυβέρνηση. Ρωτώ, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να φέρετε στο πρώτο πλάνο, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, το θέμα της εφαρμογής της οδηγίας υπηρεσιών. Το 2009 και 2010 έκανε εκθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα. Τη επέβαλε δηλαδή σε αυτό. Δεν γίνεται πλέον αυτό. Ξέρω ότι βρισκόμαστε σε διαφορετική φάση. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια όμως και γι' αυτό θέλουμε να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για το πού βρίσκεται η Ευρώπη. Να γνωρίζουμε περισσότερο γιατί δεν εφαρμόζεται συγκεκριμένα. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη accountability. Μπορείτε να επανεισαγάγετε, ε, ιδέα είναι αυτή, μπορεί να συζητήσει κανείς και άλλες ε, ιδέες. Γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες που ψάχνουν να βρουν δουλειά δεν έχουν την ευκαιρία αυτή, η οποία στο κάτω της γραφής δεν επιβαρύνει τους δημόσιους προπολογισμού. Αρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν έχω τόσο ερώτηση να κάνω, αλλά μάλλον να απαντήσω σε κάτι που αναφέρατε εσείς στην παρέμβασή σας για την πιθανότητα ενός SMA 3 στα πλαίσια μιας ψηφιακής Εσωτερική αγορά. Στη δική μα ομάδα εργασία που ζητούμε το σχετικό θέμα, ε, ξεσπάσαμε αν θέλετε σε χειροκροτήματα μόλι ακούσαμε την πρόταση. Θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα και μακάρι να μπορέσουμε να βάλουμε και σε μια σειρά όλε αυτέ τι ιδέε που έχουν ακουστεί και στη δική μα ομάδα. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σας κοινοποιήσω ότι Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας, όσο μπορεί να σας βοηθήσει η ομάδα εργασία μας. Εσάς και το γραφείο σας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το τρίτο SMA. Ναι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαρή να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα για να δούμε αν υπάρχει και άλλο χρόνο για να δώσουμε το λόγο σε άλλου αγχωρητέ. Ο κύριο Μπαρνιέ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, έτσι ώστε να υπάρξει και τρίτο γύρο, αν είναι δυνατό. η κυρία Βερνιό. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που μένουν ανοιχτά για τον τριμερή διάλογο για τα επαγγελματικά προσόντα, ένα θεμελιώδες το οποίο μπαίνει και σε άλλους τομείς της δυνατότητας μεταφοράς, της αμοιβαιότητας και της συνοχής των συστημάτων ασφαλίσεων. Συζητούσαμε πρόσφατα για τις δημόσιες προμήθειες και σχετικά με τις ασφαλίσεις που υποχρεούνται να διαθέτουν οι επιχειρήσει όταν θέλουν να μεταβούν να εργαστούν σε άλλη χώρα. Η Γενική μου Διεύθυνση αρχίζει διάλογο με τους ασφαλιστές. Έχετε δίκιο που το θέτετε αυτό το θέμα, διότι δεν αφορά μοναχά στην προστασία των καταναλωτών, αφορά την ίδια την ενιαία αγορά, διότι ασφαλώς υπάρχουν καμιά φορά πρακτικές ή και συνήθειες που οδηγούν σε διακρίσεις και επομένως εκφεύγουν το πνεύματος της ενιαίας αγοράς. Άρα, θα διεξαγάγουμε το διάλογο αυτό με τους ασφαλιστές και πιστεύω να μπορέσουμε να βρούμε ε, ε, με κοινή προσπάθεια κάποια ε, λύση ή δεμή θα χρειαστεί να αναλάβουμε δράση, δράση εμείς. Κύριε Ζουβά, εσείς, πέραν των όσων ήδη είπα σαφώς επισήμως και με δυνατή φωνή για το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έχει ούτε σήμερα ούτε αύριο την ε, ε, πρόθεση να οδηγήσει η ιδιωτικοποίηση της παροχής πόσιμου ύδατος. Να το βάλουμε. Γνωρίζω για αυτό το κείμενο αναφοράς που λέτε πράγματι να το βάλουμε επισήμως στο άρθρο πρώτο του σχετικού νομοθετήματος την εγγύηση αυτή που προσφέρουμε στους πολίτες ότι δεν υπάρχει απλώς καμία βούληση ιδιωτικοποίησης του, της παροχής του πόσιμου νερού. Σύμφωνοι λοιπόν. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Εγώ προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν ακριβέστερος και, τις, και σαφέστερος, όπως και για παράδειγμα με το βαθμολόγιο, scoreboard και, τους πίνακες, και τον πίνακα μάλλον που ε, εκδίδουμε. Χθε μάλιστα στη Γενική μου Διεύθυνση μίλησα συγκεκριμένα για τα διάφορα κεφάλαια. Τώρα θα πούμε και στις λεπτομέρειες, έτσι είναι. και η αρμόδια διευθύντρια θα μπορέσει να προσέλθει εδώ ενώπιον σας να σας εξηγήσει σημείο προς σημείο, τομέα προς τομέα, πώς θα κινηθεί η οδηγία α, περί υπηρεσιών. Σύμφωνοι να υποβάλλεται έκθεση από την Κομισιόν στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Πιο χρήσιμο μάλιστα ακόμα θα είναι αυτό, διότι για να επιτύχουμε πρέπει να κινητοποιηθούν οι ίδιες οι χώρες μέλη. Και το ίδιο και στην ε, Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής και με τη συμφωνία του Όλι Ρεν μπόρεσα να βάλω ένα κεφάλαιο για την ανταγωνιστικότητα στο ίδιο το ευρωπαϊκό εξάμεινο που δεν είναι μονάχα για κυρώσεις, λιτότητα, σκληρές κουβέντες και για τις επιχειρήσεις. Μέσα αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν πρέπει να μπουν μόνο αυτά, αλλά και η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη Αυτά λοιπόν συναποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ε, της προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τώρα, για την ε, υπόθεση αυτή της μηδενικής ανοχής. Υπενθυμίζω ότι το 2001 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης τότε είχε βάλει ένα όριο 1,5% και αυτός ο στόχος επιτεύθηκε τον Νοέμβριο του 2006, μετά από μια πενταετία από τότε δηλαδή. Το 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελών μείωσε το όριο στο 1%. Τώρα έχουμε φτάσει στο 0,6%. Άρα αποτελεί αυτό πρόοδο. Και αυτό το 0,5% θα πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος. Ευχαριστώ και τον κύριο Αρίας. Η ομάδα της οποίας προεδρεύεται κύριε κυρία Αρίας είναι σημαντική γιατί είναι ανοιχτή και στους stakeholder εγώ έχω ανάγκη από τις εργασίε τη ομάδα σας και ευχαρίστω να επανέλθω να συνεργαστούμε με την ομάδα σας που είναι ανοιχτή και συμβάλλει πραγματικά για να μπορέσουμε να προπαρασκευάσουμε το περιεχόμενο του Single Market 3 που σε μεγάλο μέρος θα αφιερωθεί και στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Well, I think the indicated... Ο Επίτροπος ε, επιτρέπει ένα ακόμη γύρο ερωτήσεων. Για να δω πόσοι συντονιστές θέλουν το λόγο. Uh, from the members. I have Mrs. Weiler, Mr. και κυρία Πέρες. Και πόσοι συντονιστές. Ναι, δεν ακούσαμε καθόλου τους πρασίνου, οπότε κυρία Ρούλερ θα πάρει το λόγο. Κέπχαρτ, κάποιος άλλος, κύριος Μπίλερ. Ρούλερ και Μπίλερ γιατί δεν ακούσαμε καθόλου τις ομάδες τους. Και μετά δώσω το λόγο στην κυρία Βάιλερ, ο κύριος Κρότσμαν και τους φιλελεύθερους. Και μετά η κυρία Κόγεν. Αποφασίστε μεταξύ σας ποιος θα θέσει την ερώτηση. Καλώς. Well, let's take everybody then. Όλοι, όλοι θα πάρετε το λόγο. Αν καταφέρετε να κάνετε την ερώτησή σας σε λιγότερο από ένα λεπτό. All right. So everybody, all the coordination... Όλοι οι συντονιστές λοιπόν θα πάρουν το λόγο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κυρία Ρούλερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και σας κύριε Επιτροπέ. Έχω ήδη προπαρασκευάσει ανακοινωθέν τύπου που επισημαίνω ότι σήμερα συμβάλλατε πολύ στην εξασφάλιση διαφάνειας. Και ιδίω για τα όσα είπατε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που ήταν η μεγάλη ανησυχία της Αυστρίας, της Γερμανίας και του Βελγίου και νομίζω ότι με τα όσα είπατε, μάλλον για τις κοινοτικές επιχειρήσεις, ε, αναφέρεται μάλλον στα νερά η κυρία Ρούλε. Με αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι και η οριζόντια δημόσια συνεργασία, η οποία καμιά φορά περνάει και τα σύνορα των χωρών μελών και ξεπερνάει και τα ε, όρια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι δημόσιες αυτές αρχές στο μέλλον θα μπορούν να συνεργάζονται στη βάση κοινών καθηκόντων και δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Αυτό ωστόσο ε, προκαλεί προβλήματα εφόσον υπάρχει συνεργασία μεταξύ μικρών κοινοτήτων και κρατών, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα ίδια κέρδη οι μικρές αυτές κοινότητες και εν ώψη του μεγάλου βάρους από το δημόσιο χρέος χρειαζόμαστε αυτή την, ε, πώς να πω, την ανταγωνιστικότητα ώστε να μπορέσουν και αυτές να ε, φτάσουν σε κάποιο εισόδημα. Ευχαριστώ πολύ για το scoreboard της τουρκικής αγοράς. Η ανακοίνωση επιτροπής ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Είπατε ότι 23 κράτη-μέλη έχουν επιτύχει το στόχο του 1% για το έλλειμμα της ε, της νομοθεσίας. Όμως υπάρχουν και κάποιες χώρες, όπως η Πολωνία χώρα μου, που δεν το επιτυχούμε αυτό το στόχο. Είναι πραγματικά ντροπή, γιατί εμείς είχαμε διοργανώσει το πρώτο φόρουμ για την ενιαία αγορά και ρωτώ τι προτίθεστε να κάνετε ως Κομισιόν για αυτά τα τέσσερα κρατημέλη που δεν έχουν επιτύχει τον στόχο. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι και ως Γάλλο ως Επίτροπο. Για το ΦΠΑ στα βιβλία. Ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Κάτι είχε υποσχεθεί η Επιτροπή και το 2013. Εμείς θα θέλαμε να μειώσουμε το ΦΠΑ στα βιβλία, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να μπορούμε να το κάνουμε. Κρότσμαν. Ευχαριστώ και εγώ για τα ξεκάθαρα λόγια σας για την οδηγία, γιατί τα όσα έχουν συμβεί στη Γερμανία είναι ένα έσχος. Έχω μία παράκληση για την διακοινοτική συνεργασία, δηλαδή μεταξύ κοινοτήτων. Έχουμε παραδείγματα μικρών κοινοτήτων που μοιράζονται ένα αυτοκίνητο σάρωθρο, αυτό που σκουπίζει τους δρόμους. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ε, ε, εγώ νομίζω ότι ο, ο Επίτροπος βρίσκεται στην ίδια αυτή γραμμή και νομίζω ότι αυτό είναι και σωστή ρύθμιση. κ. Βάιντερ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο μια παράκριση που πήγαινε λίγο μακρύτερα. Μετά τα όσα είπατε, αλλά και όσα έχετε γράψει παλαιότερα για την οδηγία παραχωρήσεων, που φαίνεται ότι κανείς δεν ανέγνωσε στη Γερμανία. Η δική μου παράκριση ήταν, αλλά και είναι, μέχρι ότου ληφθεί η τελική απόφαση, μάλλον τον Οκτώβριο δηλαδή, να κοιτάξετε με τις χώρες μέλη, οι οποίες οφείλουν και αυτές να έχουν κάποιο συμφέρον, κάποιο ενδιαφέρον να γίνει πιο αντικειμενική η συζήτηση στη Γερμανία έρχονται οι αντιπρόσωποι μα εδώ, είναι σύμφωνοι και μετά προ τα έξω στην κοινή γνώμη δεν λένε τίποτα. Να είμαστε ωστόσο και έντιμοι. Ένα μέρο τη εκστρατεία αυτή που διεξάγεται τώρα έχει και σχέση και με το γεγονό ότι ορισμένε κοινότητε βγάζουν κέρδο από την ιδιωτική χρήση του πόσιμου νερού. Εγώ είμαι αντίθετη, αλλά ορισμένε ορισμένες ε, ε, κοινότητες το πράττουν αυτό. Επίσης κύριε Επίτροπε, αν μπορείτε να μας τα πείτε αυτά και γραπτός, θα με ενδιέφερε πόσο έχει προχωρήσει η εργασία σας και η προπαρασκευή για μεταρρύθμιση της οδηγίας για τα παιχνίδια. κυρία Κόγεν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα τη μετά... Δεν κατάλαβα καλά τη μετάφραση για το τελευταίο που είπατε. Ναι, ναι, ναι, ναι, πόσο έχει προχωρήσει η εργασία σας για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τα παιχνίδια, δηλαδή τα παιχνίδια των παιδιών. Κύριε Ρικογέν, ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις στον Επίτροπο πρώτον για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς χιλιάδες ισπανικές οικογένειες υποφέρουν, καθώς εξαπατήθηκαν από τις τράπεζες. Και τα τεστ ε, ικανότητας ε, δεν φάνηκαν ικανά. Τι προτίθεστε να κάνετε για να επιλύσετε τα προβλήματα που ήδη έχουν προκύψει και να προλάβετε παρόμοιες κατάσταση Είπατε ότι στο SMA 2 για την ε, αφαιρεγγιότητα θα κάνετε κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια στη χώρα μου, καθώς χιλιάδες ισπανικές οικογένειες λόγω των συμβάσεων που έχουν υπογράψει να βρεθούν στο δρόμο. Προτίθεται η Κομισιό να προτείνει μια νέα νομοθεσία για να αποφύγουμε αυτές τις αδικίες και τις καταχρήσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις των στεγαστικών δανείων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Μπαρνιέ για τη διευκρίνηση για τις κοινωτικές επιχειρήσεις. Γιατί μου τα έχετε πει αυτά βέβαια και παλαιότερα σε συζητήσεις. Χαίρομαι που τα είπατε τώρα και δημοσία. Μπορείτε να επισημάνετε και στις υπηρεσίες σας ότι πρέπει να πράξουν το ίδιο. Είχα παρακαλέσει να με υποβάλλετε πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει σχετική διατύπωση και τα όσα μου διαβίβασαν οι υπηρεσίες σας αναγκάστηκα να τα καταφορήσω στο αρχείο, να το πω έτσι, γιατί ήταν τελείως διαφορετικά από τα όσα είχατε υποσχεθεί. Γι' αυτό και είμαι κάπως πιο συγκρατημένη τώρα με τους επένους που θα σας απίφθηνα κανονικά. Δεύτερον, εξ του συναδέλφου Μάρκ Ταραμπέλα, θα ήθελα να παρακαλέσω να επαναλάβετε την διαβεβαίωση εδώ ενώπιον μας για το, δικαί... για το δίκαιο αναθέσεων δηλαδή ότι στρατηγικά θα συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στο Συμβούλιο και όχι όπως συμβαίνει σε άλλα ντοσιέ, όχι δικά σας, όπου έχουμε δυστυχώς δει την Κομισιό να συμπαρατάσετε στο πλευρό του Συμβουλίου. Μια τέτοια διαβεβαίωση θα ήταν για μας πάρα πολύ σημαντική. Δεν θα πω άλλα γιατί δεν προλαβαίνω. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ξεκάθαρο το μετά, κύριο Σφαπ. Το τελευταίο. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα. Πρώτο, single market governance. Βεβαίω υπάρχει έλλειμμα εφαρμογή στι χώρε μέλη και είναι σημαντικό δείκτη αυτό. Το μέγα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τόσο η εφαρμογή, όσο η εφαρμογή στην καθημερινή ζωή, όχι μεταφορά δηλαδή στα δίκαια, αλλά η εφαρμογή στην καθημερινή πράξη. Άρα εδώ χρειάζεται διαφάνεια. Δεύτερο, η, πρωτοβουλία πολιτών δικαίωμα στο νερό, right to water, νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο χρειάζεται πολιτική απάντηση από την Κομισιόν, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή που εξήγησε προηγουμένως ο εισηγητής μας κ. Ζουβά. Δεν μπορεί όμως να μείνει εκκρεμής, διότι κάποια στιγμή θα μας στάσει η πρωτοβουλία πολιτών με τις υπογραφές όσο το δυνατόν συντομότερο λοιπόν ώστε να μπορέσει να συζητηθεί και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα για το Single Market Act 3 έχουμε ταυτόχρονα τέσσερις μεγάλες οδηγίες που πρέπει να μπουν στους τριμερείς διαλόγους. Η επιβάρυνση για τους συναδέλφους μου είναι τεράστια, το φόρτο, εργασίας δηλαδή. Γι' αυτό παρακαλώ ασφαλώς να κρατήσουμε τον στόχο του Single Market Τρία, να μην κατακαιρματιστούν όμως οι προσπάθειές μας ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Μπανιέ, να απαντήσει και πάλι. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλα, μάλιστα, θεωρώ ότι η οριζόντια συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική και θέλουμε να τη διασφαλίσουμε. Γι' αυτό ακριβώς συμπεριλάβαμε την οριζόντια συνεργασία μεταξύ Δήμων, χωρίς να είναι απαραίτητα Πολλές φορές είναι και διαμεθοριακή. Συμπεριλάβουμε λοιπόν αυτή την πτυχή ε, στις προτάσεις για τις δημόσιες προμήθειες ε, και τις ε, παραχωρήσεις. Ίσως να μην αρκεί, όμως η αρχή εξακολουθεί να ισχύει και πρόκειται για πραγματική συνεργασία με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όμως θέλουμε να ενισχύσουμε την οριζόντια αυτή συνεργασία, ιδιαίτερα στο κείμενο για τις παραχωρήσεις και θα εξακολουθήσω να συνεργάζομαι με τον εισηγητή για αυτό το ζήτημα. Ανέφερα και προηγουμένω τι συμβαίνει με τα Stadtwerke και του όμορου Δήμου. Ότι δηλαδή θα πρέπει να χειρίζονται και τα δημόσια οικονομικά με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και βεβαίω θα προσπαθήσουμε να βρούμε και ένα πιο ξεκαθαρό τρόπο. κύριο, Βιλάν, βεβαίω και ο απολογισμό ε, τη ε, μεταφορά στην εθνική νομοθεσία που μόλι δημοσιεύσαμε πράγματι δείχνει ότι δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. για ορισμένε χώρε, όμω ε, πρέπει να ενθαρρύνουμε τι χώρε που παρουσιάζουν καθυστέρηση να προχωρήσουν. Και σε ό,τι αφορά αυτή την εικόνα, πρέπει να σα πω ότι ε, διεξάγουμε και νέου διαλόγου με τι κυβερνήσει ε, των χωρών ε, που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Όπω για παράδειγμα με την πολωνική κυβέρνηση με τι επόμενε εβδομάδε. Γιατί δεν είναι μόνο να του κάνουμε παρατήρηση. Μπορούμε να κάνουμε διαδικασίε επί παραβάση. υπάρχει και η μηδενική ανοχή, όμω Έχω συναντήσει όλους τους υπαλλήλους που έχουν αναλάβει ε, την ε, οδηγία υπηρεσιών για να αναλάβουν προσωπικά αυτή την σωστή εφαρμογή της ε, οδηγίας. Πρέπει δηλαδή να έχουν και μια θετική γνώμη των Βρυξελών. Δεν έχω κατά νου το σημείο για τον ΦΠΑ. Όμως ε, σίγουρα θα το διευκρινίσουμε και μαζί. Ενδεχομένως ε, με τον ε, συνάδελφο που έδειξε το ζήτημα. Κύριε Κρόιτσμαν, σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε, για τις διευκρινίσεις. Και πάλι είμαι πολιτικός, όπως είστε κι εσείς. Και δεν μεταράζει ταράζει αυτός ο δημόσιο διάλογος, αυτές οι αιτήσει, όταν γίνονται σωστοί ισχυρισμοί. Επισήμως σας ανέφερα προηγουμένως ε, την προσωπική μου πεποίθηση αλλά και της Επιτροπής ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον να υπάρξει ιδιωτικοποίηση ε, των υπηρεσιών ύδατος. Αλλά κάποιος προηγουμένως είπε ναι, αλλά οι υπηρεσίες ε, δεν έκαναν αυτό που είπα. Ήδη έχει σημειωθεί μια πρόοδος ε, που δεν υπήρχε προηγουμένως ε, στο κείμενο και σας άκουσα λοιπόν, άκουσα και τον εισηγητή. Άκουσα τον κύριο Κρόιτσμαν, τον κύριο Σουάμπ. Γι' αυτό και θεωρώ ότι προς διευκρίνηση θα πρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις κακές ερμηνείες. Έχω συμπεριλάβει λοιπόν μια νέα πρόταση που δεν υπήρχε στο κείμενο, αλλά με τα χαρά να πω στι υπηρεσίε μου να έρθω σε επαφή μαζί σα για πιο συγκεκριμένα στοιχεία για να είστε και σίγουροι ότι αυτό που λέει ο Επίτροπος αντικατοπτρίζεται και στα όσα αναφέρονται, σε αυτά που αναφέρουν οι, οι υπηρεσίες. Κυρία Βάιλερ. Για αυτή τη σημαντική πρόοδο που, κατά τη γνώμη μου, που έχει επιτευχθεί, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ε, στη Γερμανία, στην Αυστρία, Γι' αυτό που επανέλαβα και προηγουμένως ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ιδιωτικοποίησης. Ε, πράγματι, θεωρώ ότι θα πρέπει να, κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων, να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο πλαίσιο ε, για τις παραχωρήσεις, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Σας υπενθυμίζω ότι η έλλειψη τέτοιων κανόνων μπορεί να αποβεί σε βάρος ε, των ε, πολιτών, να υπάρξουν περιπτώσεις διαφθοράς, διακρίσεων. Βρισκόμαστε στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και έτσι έχουμε μια τέτοια ευθύνη, χωρίς να ε, θέσουμε ανεφιβόλο το δημόσιο χαρακτήρα αγαθών όπως το νερό, αλλά και την ελευθερία και την, ε, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των τοπικών αρχών. Οι ίδιες λοιπόν αποφασίζουν. Μετά αναφέρθηκε η πρόταση ε, των ε, στεγαστικών ε, δανείων που υιοθετήθηκε στις 31 Μαρτίου και η Ιρλανδική Προεδρία ασχολείται με αυτό το θέμα όπως και εγώ. Καθώς είναι μία από τις πτυχές της κρίσης την οποία δερχόμεθα. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τα στεγαστικά δάνεια. Και ο εισηγητής ε, είναι ιδιαίτερα δραστήριος ε, σε αυτό το θέμα. Εδώ να υπογραμμίσω μια μικρή παρανόηση. Εγώ ως Επίτροπος ε, καταρτίζω κείμενα που μπορεί να απαντούν ε, σε προκλήσεις της κρίσης ή ε, να ενεργούν προκαταβολικά ε, για ορισμένα προβλήματα. Μπορώ να, λοιπόν να πω ένα από το Κοινοβουλίο ότι κανένας κλάδος ή φορέας δεν πρόκειται να ξεφύγει από ε, τους κανόνες της ε, ενιαίας αγοράς. 28 νόμους έχω προτείνει μέσα σε τρία χρόνια και οι περισσότεροι από αυτοί εγκρίθηκαν. Μιλάμε για 610 εκατομμύρια δολάρια που ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία που τα συζητήσαμε τα τελευταία χρόνια και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα στις ε, είπα, ζήτησα από τους Αμερικανούς και από τους, τα υπόλοιπα μέλη του G20 να κάνουν το ίδιο. Επομένως έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον ε, σε ό,τι αφορά τους, ε, τον έλεγχο των τραπεζών, ε, την ανακεφαλοποίηση. Ούτως ώστε οι τραπεζίτες πράγματι και η δράση τους μάλλον να ποινικοποιείται όταν υπάρχει κατάχρηση εξουσίας, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα διαφθοράς και να υπάρχουν και ποινικέ κυρώσει όταν είναι, ε, τα, τα αντικείμενα αυτά είναι πράγματι πιο σοβαρά. Και βεβαίω να λαμβάνουμε δράση και για να στηρίξουμε τους πολίτες ε, που βρίσκονται εν μέσω κρίση αυτή τη στιγμή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Well, thank you very much as always. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όπως πάντοτε, 15 ερωτήσει. Παγκόσμιο ρεκόρ. Θα συνεχίσουμε πέσει στις επαφές μας. Χαιρόμαι ιδιαίτερα για τη σημερινή σας πρωινή παρουσία εδώ. Thank you. Did you see that? you So I ask anybody who's not staying for the next two presentations... If... Όποιος ε, δεν θέλει, όσοι θέλετε να μην παρακολουθείς τις επόμενες ε, παρουσιάσεις, να φύγετε σιωπηρά. Παρακαλώ πολύ. Έχουμε ακόμα δύο παρουσιάσεις. Θα ξεκινήσουμε συζητώντα ε, την πρόταση της κυρίας Βάιλερ για τον εξοπλισμό. Μπορεί να μην υπάρχει χρόνος ιδιαίτερα για πολλές ερωτήσεις, αλλά θα υπάρξει μια πρώτη παρουσίαση και έπειτα υπάρχει μια δεύτερη πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αφορά το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Σας ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους γιατί κράτησαν τον ελάχιστο χρόνο ως τώρα στην αγορεύσή τους, ώστε να τίθενται ερωτήσεις και να μπορούν ε, να ακούγονται και απαντήσεις. Κύριε ήσασταν ο μόνο που δεν τα καταφέρατε, ελπίζω να μην μου κρατάτε κακία. Μα εντάξει δεν με ακούτε ούτω ή άλλω τι λέω, οπότε δεν πειράζει. Σας ζητούσα συγγνώμη. Απλά ζητούσα συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να σας ε, λάβουμε υπόψη και να κάνετε το ερώτημά σα. Την επόμενη φορά όμως θα σας ξεχάσω. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά θέλω να χαιρετήσω εδώ στο βήμα και τον ε, κύριο Ζηρά της αρμόδιας μονάδας ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν γνωστό στην Επιτροπή μας και σε μένα γιατί δουλεύει για έναν φάκελο που αφορά τα, τα σκάφη αναψυχής. Και βλέπω ότι μεγάλη ευκολία περάσατε από τα σκάφη αναψυχής στον ραδιοξοπλισμό. Μια νέα πρόταση ουσιαστικά ε, αναθεώρηση της νομοθεσίας, η συγγήτρια κυρία Βάιλερ και σύμφωνα με ό,τι συμφωνήσαμε στους τονιστές ε, το 2009, καλέσαμε μια, την Κομισιόν για μια μελέτη τεκτύπου. Οπότε θα σας δώσω αμέσω το λόγο και αν καταφέρετε να μην ξεπεράσω δεκάλεπτο, θα έχουμε, σχόλια, θα έχουμε λίγο χρόνο για ένα-δύο σχόλια ακόμα και ε, μετά κύριε Βάλερ θα πρέπει να έρθει σε επαφή με του σκιώδε, όπω και εγώ θέλω σκιώδες. Κύριο Βαντεκάπ επίσης άλλο σκιώδες. Δύο σκιώδες είναι παρόντο αυτή τη στιγμή. Α, και ο κύριο Μάντερ. Τρει. Έχουμε λοιπόν ε, την αφρόκρεμα των ε, σκιωδών. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια, κύριε Ζωράρη, για την οδηγία του ροδιοξοπλισμού. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι τιμή και χαρά μου να παραβρίσκομαι σε εργασίες της Επιτροπής σας και να σας πληροφορώ για οποιοδήποτε θέμα θέλετε κάποιες διευκρινήσεις. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την επανεξέταση της γνωστής οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού και τερματικά του τηλεπικοινωνιών. Μιλούμε δηλαδή για έναν τομέα, πρώτα απ' όλα θα για την πλέον τύπου και για την πρόταση. Εδώ μιλάμε για έναν τομέα που έχει περίπου 80 δις παραγωγής, μια μικρή μείωση αντιμετώπισε λόγω της κρίσης όπως και άλλη βιομηχανική κλάδη. Και υπάρχει ένα ε, έλλειμμα περίπου 7 δις το χρόνο. Η οδηγία αυτή είναι, ακολουθεί μια νέα προσέγγιση, δηλαδή ορίζει τις ουσιώδεις απαιτήσει και έπειτα τις διαδικασίες για τον καθορισμό αναρμονισμένων προτύπων, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της οδηγίας, όπως και την ευθύνη του κατασκευαστή, του ε, διανομέα και των αρχών παρακολούθησης υποπτήρες αγοράς. Οι συζητήσεις που είχαμε στα πλαίσια της κείμενης οδηγίας μας έδειξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πολλά τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε, όμως απαιτούνται κάποιες προσαρμογές για να είναι καλύτερη η νομοθεσία ώστε να εφαρμόζεται και καλύτερα. Η διαδικασία ξεκίνησε το 2007 μια δημόσια διαβούλευση για τα θέματα που χρήζουν επανεξέτασης και μετά με τι συζητήσει με του εκπροσώπου των κρατών μελών, του εκπροσώπου κατασκευαστών, καταναλωτών, φορέων κοινοποίηση, προτύπων, και ξεκίνησε και η διαδικασία η επίσημη το 2010 με μια νέα δημόσια διαβούλευση το και το 2010 ώστε να εξετάσουμε τις δυνατότητες που υπήρχαν στο τραπέζι και τέλος υιοθετήθηκε η πρόταση τον Οκτώβριο του 2012 από την Επιτροπή. Άρα, ποια είναι τα βασικά ζητήματα εν προκειμένου. Πρώτα απ' όλα το πείσαμε ένα χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης πολλές εκστρατείες που έγιναν για να δούμε ποιο το επίπεδο της συμμόρφωσης και ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος και τις περίοδους χρόνου, τα επίπεδα ουσιαστικής συμμόρφωσης ήταν ανάμεσα στο 28% και 56%. Άρα, μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης. και αυτό σχετίζεται και με τα θέματα της συχνηλασιμότητας των προϊόντων. Διευκρινήσεις που χρειάζονται δηλαδή για τον ορισμό των ίδιων των προϊόντων. Όταν τα επίπεδα συμμόρφωσης είναι τόσα χαμηλά, αυτό τι δείχνει αθέμεντο αγωνισμό αυτών που δεν συμμορφούνται με τον νόμο και αυτό είναι εις βάρος όσων συμμορφούνται με τον νόμο. Και δημιουργεί και σοβαρό πρόβλημα και στην αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος. Άλλος τομέας ε, που, στον οποίο πρέπει να σκέψουμε και να δούμε αφορά την ε, διευκρίνηση κάποιων διατάξεων. Μία από τις που ζητήθηκε αφορά τους παραλήπτες. Παραλήπτες που είναι στο πεδίο εφαρμογή οδηγίας. Και ποιοι είναι μέσα και ποιοι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή. Ένα ζήτημα που φάνηκε να δημιουργεί προβλήματα στην ε, εφαρμογή της νομοθεσίας, διότι υπάρχει και μια άλλη οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και εκεί οι ουσιώδες απαιτήσει που πρέπει να εφαρμόζονται είναι πια από τις δύο οδηγίες. Εκεί υπήρχε μια σύγχυση και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το πεδίο εφαρμογής για την αναθεωρημένη αυτή οδηγία θα πρέπει να αφορά μόνο τον αραδιοεξοπλισμό με δυνατότητες εκπομπής. Άρα δηλαδή η, τα σημεία εκπομπής είναι στο πεδίο εφαρμογής ή αποδέκτες όμως, οι λήπτες δεν είναι ε, εντός η δέκτας δεν είναι ε, εντός. Και τέλος ένα άλλο σημείο που ετέθη από πολλούς συμμετέχοντες συζήτηση ήταν ότι η κείμενη οδηγία δεν προβλέπει διατάξεις που μπορούν να εγγυηθούν τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στον αδεξοπλισμό με τα ένας τομέας που εγείρει πολλά ζητήματα και ερωτήσει σχετικά είναι οι φορτιστές κινητών τηλεφώνων. Κάτι που δεν προβλεπόταν, δεν είχε συμπεριληφθεί στην προηγούμενη Και Τέλος, ένας ακόμη τομέας ε, που έγινε ερωτηματικά ήταν πιθανά ρυθμιστικά εμπόδια για την είσοδο νέων ε, εξαρτημάτων νέου εξοπλισμού στην αγορά. Και μετά από συζητήσει καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτά είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας και συνδέονται πιο πολύ με την εναρμόνιση του φάσματος, κατανομή ε, και αδειοδότηση ε, του φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι μια άλλη διαδικασία. Και αφορά μια άλλη νομοθετική πράξη. Η μελέτη λοιπόν αντικτύπου, οι στόχοι αν θέλετε που εντοπίστηκαν, να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα να βελτιώσουμε την εφαρμογή, όπως είπα, και τη συμμόρφωση με την οδηγία. Δεύτερο στόχος, να υπάρχει μία στερεά νομική βάση που να επιτρέπει την εφαρμογή των ουσιοδών ε, απαιτήσεων και ο τρίτος στόχος είναι πώς να άρουμε τα ρυθμιστικά εμπόδια για την πρόσβαση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων ε, ραδιοξοπλισμού. Σε ό,τι αφορά το πρώτο στόχο, η επιλογή που επιλέξαμε ήταν αυτή που μιλάει για πλήρη ευθυγράμμιση της οδηγίας με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. και που θα μας επιτρέψει να εισάγουμε απαιτήσει καταχώρησης για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες εξοπλισμού όταν δεν επιτυγχάνεται ψηλό επίπεδο συμμόρφωση. Ε, δύο λόγια μόνο για αυτό το θέμα του Μητρώου, της καταχώρηση, γιατί αυτό το ζητά η Κομισιόν με πράξη καταξιοδότηση η Κομισιόν και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι ε, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτόματη καταχώρηση εξοπλισμού. Αυτό που θέλουμε είναι οι αρχές αποπτήρες αγοράς να εντοπίσουν κατά πόσον υπάρχει εξοπλισμός που συστηματικά δεν συμμορφούνται με την νομοθεσία και αν υπάρχει κάτι τέτοιο και αν αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη πρέπει να αναλυφθεί δράση. Για παράδειγμα, τα walkie-talkies σε ένα νοσοκομείο που μπορεί να παρεμβαίνουν στον ιατρικό εξοπλισμό. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Για το δεύτερο στόχο, ο στόχος Β. Προτείνουμε λοιπόν στην Αθημένη Οδηγία την ε, διευκρίνηση, την επεξήγηση κάποιων ε, διατάξεων και την απλούστευση των διοικητικών υποχρεώσεων. και ζητείται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δοθεί η εξουσία στην Κομισιόν ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της οδηγίας σε κάποιους τομείς, τομείς ε, όπου νέος εξοπλισμός ε, λειτουργεί με ένα λογισμικό τέτοιο το οποίο ε, έχει καθοριστικό παράγοντα στην χρήση αυτού του εξοπλισμού. Και ότι εδώ εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογή όλη η κατηγορία των πομπών. Έπειτα, κατηγορία Γ. Κάτι που δεν αφορά το πεδίο εφαρμογή. Τι δεν αφορά το πεδίο εφαρμογή, τι είναι εκτό. Και προτείνεται να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σημείο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται τα αιτήματα για πειραματικές άδειε για τη χρήση ραδιοξοπλισμού και ένα σχέδιο δράση για τη βελτίωση των εργασία ανάμεσα στι ρυθμιστικέ αρχέ φορείς κοινοποίηση και προτύπων. Θα περάσω τώρα στην νομοθετική πρόταση. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, να δούμε τις κύριες αλλαγές. Ε, η πρώτη και βασική και σημαντική αλλαγή είναι η ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τους ορισμούς, τις υποχρεώσεις των ε, εμπόρων ε, τα έντυπα για την αξιολόγηση συμμόρφωσης, υποχρεώσει κοινοποίηση τη συμμόρφωσης και σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, ένα νέο ορισμό για τον ραδιοξοπλισμό που να συμπεριλαμβάνει μόνο τον εξοπλισμό εκείνο που σκοπίμως ε, μεταδίδει σήμα και χρησιμοποιεί το ραδιοφάσμα. Ο επόμενος ε, τομέας ε, τη οδηγία που στι αλλαγέ. Βλέπετε στο άρθρο 3 προβλέπετε η δυνατότητα νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την λειτουργικότητα των αξεσουάρτων ε, αξεσουάρ των προϊόντων αυτών. Έπειτα βλέπετε ότι μιλάμε για δυνατότητα καταχώρησης και κάποιες διευκρινήσεις για τη σχέση ανάμεσα σε αυτή την οδηγία και την ομοθεσία σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος. Όπως επίσης την απλούστευση των διοικητικών υποχρεώσεων. Τέλος. Ευθυγράμμιση με τη συνθήκη και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτελεστικές εξουσίες που ζητάει η Κομισιόν βάσει όσων προβλέπεται στο άρθρο 8.3 και του 19 ε, ναι, ε, και πράξη καταξιοδότηση σύμφωνα με ό,τι προβλέπει το άρθρο 2 παραγράφος 3 προσαρμογή τεχνική πρόοδο δηλαδή άρθρο 3.3 κατηγορίες ε, εξοπλισμού που θα πρέπει να ταυτοποιούνται και αφορούν ουσιώδεις ε, υποχρεώσεις και το 4.2 διατάξεις για τη συμμόρφωση του λογισμικού α, που το οποίο φέρουν ε, αυτά τα προϊόντα ραδιοξοπλισμού και το άρθρο 5.2 για την καταχώρηση του ραδιοεξοπλισμού για σημερινές κατηγορίες. Ε, συνοπτικά αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που μας απασχόλησαν και αυτές είναι οι βασικές διαφορές που προτείνουμε σε σχέση με την κείμενη οδηγία. Και βεβαίως είμαστε στη θέση σας να σας δώσουμε και πιο πολλές εξηγήσεις, πιο πολλές λεπτομέρειες για οποιοδήποτε σημείο της πρότασης. Ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, μεν μιλήσατε κάπως περισσότερο, αλλά καλά τα είπατε γιατί έτσι μας βοηθήσατε. Τώρα, αν θέλουν η κυρία Βάιλερ και οι σκιώδεις εισηγητέ μπορούν να παρέμβουν. Ας ακούσουμε κάποια πρώτη αντίδραση από την κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω τυπικά πώς θα προχωρήσει η υπόθεση αυτή, διότι η πρώτη μεγάλη συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων ε, των πολιτικών ομάδων για τέτοια συζήτηση δεν υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να γίνει όμως όταν σήμερα να συζητήσουμε δηλαδή διεξοδικότερα, διότι πολιτικά ε, δεν είναι αμφιλογόμενη η οδηγία, χωρίς ωστόσο να είναι και μόνο τεχνικού χαρακτήρα, διότι για πολίτες και καταναλωτές είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πολλές επιπτώσεις περί των οποίων πολλοί δεν έχουν ξεκάθαρη ιδέα. Γι' αυτό και ευχαριστώ την Κομισιόν για την σύντομη σύνοψη που υπέβαλε. Για τις και τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το θέμα, συνιστώ την ε, σύνοψη της μελέτης επιπτώσεων, που και αυτή είναι πολύ χρήσιμη για την συζήτησή μας. Οι διάφορες επιλογές α4 έως c10 δεν μας βοηθούν πολύ. Εμείς θα πρέπει να κρίνουμε πολιτικά ποιες είναι οι ευνοϊκότερες. Βέβαια, καλά είναι να απλουστεύεται η φυστάμενη νομοθεσία, να προσαρμόζεται στις ε, τρέχουσες συνθήκες και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό άλλωστε γίνεται στην περίπτωση αυτή. Για μένα και την πολιτική μου ομάδα είναι σημαντικό η προστασία των καταναλωτών να τεθεί στο προσκήνιο. Ειδικά δε, επειδή κυκλοφορούν στην αγορά πολλά προϊόντα τα οποία δεν είναι σύμμορφα, γι' αυτό είναι σημαντικό να περιληφθούν και άλλα πρότυπα. Είναι σωστό που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλευτεί με οργανώσεις προστασίας καταναλωτών και για το λεγόμενο follow-up. Εγώ θα ήθελα και για το πρώτο έγγραφο να είχαμε την έκθεση του εντεταλμένου την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ελπίζω να την έχουμε τις επόμενες ημέρες. Πέραν της προστασίας των καταναλωτών, για μας σημαντική είναι και η πρακτική εφαρμογή. Να είναι όντως δηλαδή απλούστευση. Είδα ορισμένες διοικητικές διατάξεις πολύ αμφισβητήσιμες και περίπλοκους κανόνες στο παρελθόν που θεωρώ ότι είναι απα... απολύτως περιτές. Τέλος πάντων διδασκόμαστε από αυτά. Οι δύο μεγάλοι τομείς που πρέπει να μας απασχολήσουν διεξοδικότερα αφενός το λεγόμενο scope, το πεδίο εφαρμογή δηλαδή, όπου ακόμα εμεί, αλλά και εγώ προσωπικά δεν έχω καταλήξει μέχρι πού θα φτάσουμε και δεύτερο η καταχώρηση. Καλά που δεν θα γίνεται αυτόματα, είναι καλό αυτό, αλλά πρέπει να ξαναθέσουμε το θέμα. Γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν ορισμένες ορισμένοι οικονομικοί σύνδεσμοι οι οποίοι προτάσουν αυτή την καταχώρηση χωρίς να θέλουν να, ε, προ, ε, να, συνεισφέρουν κανένα άλλο ε, δεδομένο. Τώρα για την κατεξουσιοδότηση πράξη. Εμείς βάζουμε τρία ερωτηματικά από πίσω. Όχι ότι είμαστε καταρχήν αντίθετοι, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε τι είδους εξουσιοδότηση θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις χώρες μέλη για την περαιτέρω εξέταση. για την υποχρέωση μεταφράσεως της Declaration of Conformity και για την ιχνηλασιμότητά ε, της, αυτή πρέπει να συζητηθεί εδώ μεταξύ μας, καθώς επίσης και η διασφάλιση ότι θα υπάρχει μια συνεκτικότητα και μεταξύ των άλλων οδηγιών, όπως για παράδειγμα της κυρίας Ρόιτοβα που συντάσσει έκθεση που άπτεται και του το του θέματος. Να δούμε λοιπόν ή επίσης η οδηγία για τις ε, συχνότητες των τηλεπικοινωνιών. Επίσης και, ε, και αυτή πρέπει να δούμε που εντάσσεται. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Το λεγόμενο feedback επιτόπου είναι σημαντικό. Δεν είναι γραφειοκρατία. Οι χρήστες επιτόπου γνωρίζουν καλύτερα και τη λειτουργή και που εντοπίζουν τα ελλείμματα και από πριν αλλά και με τη νέα οδηγία. Εν τέλει θεωρώ την υπόθεση αυτή λογική πολιτικά θα μας ωφελήσει αν πούμε ότι μπορούμε να πιέσουμε τους κατασκευαστές να φτιάξουν ενιαίας μορφής φορτιστές, γιατί ακούω την φήμη ότι ορισμένοι κατασκευαστές αποχωρούν από τη συμφωνία. Προσπαθούν δηλαδή να μας πιέσουν. Υπάρχουν κατασκευαστικές εταιρείες που φτιάχνουν για παράδειγμα κινητά τηλέφωνα και κάθε φορά με διαφορετικούς φορτιστές επίσης και η δυνατότητα για τους καταναλωτές και για μικρής εμβέλειας και μικρής εμβέλειας συχνότητες να μπορούν να χρησιμοποιούν πόσο υπάρχουν τέτοιες και άλλα ηλεκτρονικά μηχανήματα που διαθέτουν όπως για παράδειγμα ακόμα και τις ηλεκτρικές τους οδοντόβουρσες. Αυτά για την ώρα. Περιμένω ακόμα να βγει αυτή η οδοντόβουρτσα με το τηλεχειριστήριο. Κύριε Βαντακάμ, κύριε Μάντερς. Μιλήστε για την αρχή που σας είναι τόσο σημαντική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατανοώ ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι εδώ έχουμε ένα από τα κοσμήματα, πιο πολύτιμα κομμάτια της ε, ενιαίας αγοράς. Όμως ε, εδώ με την υφιστάμενη οδηγία που προκύπτει και από την εξόλυση δικτύπου ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί, λυπούμε λίγο γιατί έχουμε πολύ χαμηλές ε, βαθμολογίες και μπορούμε να εξετήσουμε την έκθεση της κυρίας Βάιλερ για να τεθούν κάποια εύλογα ερωτήματα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον ε, η κατάσταση στη σημερινή αγορά. Ε, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις κυρία Βάιλερ. Τρεις μόνο να ε, αφαιρέσω. Πρώτον το σύστημα καταχώρησης και εκείνη αναφέρθηκε σε αυτό. Μήπως υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας περαιτέρω γραφειοκρατίας σε σχέση με τα αποτελέσματα της καταχώρησης. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο, τα προϊόντα από τρίτες χώρες. Όπως προτείνεται αυτή τη στιγμή στο άρθρο 6, δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο σαφές με ποιον τρόπο αυτά τα προϊόντα από τρίτες χώρες με ποιον τρόπο τίθεται ρητά ε, στο πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Και τέλος, για τις καταξιδότηση πράξεις και για τις ε, εφαρμοστικές πράξεις, για μας αυτά θα μπορούσαν να απλωστευθούν περαιτέρω, για να, να δούμε πότε ακριβώς αρμόζει να μιλάμε για ταξιδότηση και πότε για ε, εκτελεστικές. Όπως στο άρθρο 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Ευχαριστώ. Ε, κύριος Μανέρς. Ευχαριστώ. Χθες ε, το απόγευμα με ορίσατε ως ε, σκιώδη συγητή, δεν ε, προετοιμάστηκα, υπήρξε έλλειψη ενδιαφέροντος αυτό το φάκελο και μετά ως συντονιστής κάποιος γίνεται ουσιαστικά ένα σκουπιδεντενικές. Όμως γνωρίζω τον συνάδελφο που το έχει αναλάβει και πολύ καιρό και έχω ένα ερώτημα σε ό,τι φορά την τυποποίηση των ε, χρεώσεων, ο, κύριος, ο Πίτροπος Σαϊτατζάνη, ε, των φορτιστών, συγγνώμη. Αυτή είναι η οδηγία όπου μπορεί να μπει αυτό το σημείο ή η Επιτροπή θα προτείνει κάτι άλλο. Γιατί ανακοινώθηκε ότι είτε θα πρόκειται για ένα θελοντικό σύστημα όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, είτε θα προτείνει κάποια νομοθεσία που θα τους υποχρεώνει. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ε, για ερωτήσει αυτή τη στιγμή, εκτός και αν ο κ. Τζιράου μπορεί να, κάνει, να απαντήσει μέσα σε ένα λεπτό, αλλά σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό. Σίγουρα η κυρία Βάιλερ θα συγκεντρώσει όλους τους κοιόδης σε το συντομότερο δυνατόν και, έτσι ίσως ο κύριος Ζηράου μπορεί να παρευρεθεί σε μία ε, συνάντηση των σκιωδών και να τα συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες εκεί. Έχετε σύντομες καταληκτικές παρατηρήσεις γιατί έχουμε και άλλη παρουσίαση στη συνέχεια. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Δεν σαν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα ακόμη, αλλά εμείς είμαστε διάθεσοι να σας εξηγήσουμε όταν ε, προκύψει θέμα, να εξηγήσουμε οτιδήποτε για τους ε, φορτιστές των κινητών τηλεφώνων. Ναι, στην οδηγία αυτή ανοίγει πλέον νομική βάση για να παρουσιάσουμε μια πρόταση για αυτό το τομέα, αν ποτέ είναι αναγκαίο. Ευχαριστώ. Okay, well, thank you very much indeed for doing that. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η έκθεση της κυρίας Βάιλερ θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική έκθεση έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα στις τουρκικές αγοράς. που το απασχολεί εδώ και καιρό και η δική μου συμβολή ως σκιώθεση είναι ότι θα πρέπει να δούμε και άλλα θέματα όπως είναι η προσπελασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες όπως έγινε στην οδηγία με τις καθολικές υπηρεσίες. Και υπήρχε σύνδεση ανάμεσα σε εκείνη την οδηγία και την προσπελασιμότητα των ατόμων σε μειονεκτική θέση και άτομα με ειδικέ ανάγκε. Είναι κάτι λοιπόν που θα θέλαμε να δούμε και εδώ. Σα ευχαριστώ όλου. Προχωρούμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα το πρωί. Λάβαμε μια παρουσίαση για τη δική μας μελέτη αντικτύπου που έγινε από τη δική μας αρμόδια μονάδα, όπως και την μελέτη, ε, την μελέτη της αντικτύπου που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Η ομάδα που δούλευε αυτό το θέμα, Πίτερ Μάγερ και Κεφάρτο, κ. Κρόιτσμαν, κ. Φόξ δεν νομίζω ότι είναι εδώ, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία του Γιώργου Πολών. Κ. Μπαλόν, δεν ξέρω ποιο θα μα παρουσιάσει τα αποτελέσματα τη έρευνα. Κυρία Παλόν, ιδιαίτερα γνωστή στην Επιτροπή μας, Θα έχετε εργαστεί σκληρά και για πολλά χρόνια στη γραμματεία της Επιτροπής και τώρα είστε επικεφαλής της μονάδας αξιολόγησης. Θα σας δώσω το λόγο να μας παρουσιάσετε τα βασικά συμπεράσματα και αν ε, συμφωνεί και ο εισηγητής, να, η εισηγήτρια μάλλον, πρώτα να ακούσουμε αυτή την παρουσίαση. Και πολλά άλλα δεν θα προλάβουμε να κάνουμε το πρωί. Θα μας πούν όμως ο εισηγητής και σκιώδας τι θα κάνουμε. Κυρία Παλών, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τη δουλειά που κάναμε Την ίδια παρουσίαση την κάναμε και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα και για εσάς. Γιατί η ΙΜΚΟ ήταν η Επιτροπή που μας ζήτησε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να κάνουμε ένα είδος ε, διάγνωσης ε, ενό διαγνωστικού, αν θέλετε, ελέγχου τη υγεία ε, και στον τομέα αυτό του δικαίου των πολίσεων. Ο σκοπό αυτή τη άσκηση είναι να δούμε κατά πόσον υπάρχει τα αντικτύπου αντικτύπωτη Κομισιόν ώστε να μπορούν τα μέλη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αργότερα να αποσπάσουν από αυτή τη μελέτη χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να μπορούν να κρίνουν με βάση συγκεκριμένα δεδομένα. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και θα σας παραπέμψω για τις λεπτομέρειες ε, στο κείμενό μας. Και μάλιστα να σας πω ότι έχουμε δημοσιεύσει δύο κείμενα. Από τη μία έχουμε τη δική μας λεπτομερή εκτίμηση και από την άλλη υπάρχει ένα ερευνητικό έγγραφο από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, τον καθηγητή Κόβατς του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνα, στον οποίο θέσαμε κάποια ερωτήματα για πολύ τεχνικά ζητήματα και τη δουλειά του τη χρησιμοποιήσαμε ως βάση για τη δική μας δουλειά. Βλέπετε λοιπόν ότι δημοσίευσαμε δύο χωριστά κείμενα και που επί της πρέπει να είναι, στο, να μπροστά σας. Λοιπόν, τα συμπεράσματά μας. Συνολικά μπορώ να πω ότι αν διαβάσετε μελέτη τύπου, είναι μία από τις καλύτερες ε, που έχουμε δει ποτέ από την Επιτροπή με όλα τα προβλήματα και τις αδυναμίες που θα θίξω σε λίγο. Αν τη δείτε λοιπόν αυτή τη μελέτη και τη συγκρίνετε με τις κατευθύνες γραμμές της Κομισιόν όπου ορίζεται η μεθολογία για τον τρόπο που εκπονούνται οι μελέτες αντικτύπου, ε, δεν είναι και κακογραμμένη. Ε, ε, έχει ένα σοβα... σαφές πρόβλημα α, στο πώς γίνεται, στο θέμα των ορισμών, και παρότι κάποια πράγματα είναι σπάνια, πρέπει να το πούμε ότι ποσοτικοποιεί ε, το κόστος και το όφελος ε, της πρότασης. Να, ένα από τα υπέρ της μελέτης αντικτύπου. Αλλά ταυτόχρονα αυτό δείχνει και την αδυναμία της. Γιατί η αδυναμία σε αυτή τη μελέτη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Κομισιόν χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα ή μη διαθέσιμα σε αυτή την περίπτωση δεδομένα για να οδηγηθεί σε ποσοτικά συμπεράσματα για το κόστος και το όφελο. Θα μπω σε κάποιε λεπτομέρειε σε αυτό το σημείο, γιατί είναι και το κεντρικό στοιχείο τη συζήτηση. Η βασική έννοια που χρησιμοποιεί στη μελέτη αντικτύπου είναι το κόστος των συναλλαγών, που ορίζονται στη μελέτη αντικτύπου ως περιορισμένα στις δαπάνες εκείνες που συνδέονται συγκεκριμένα με το διασυνοριακό εμπόριο και συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση απορρέουν από τις διαφορές στο ε, ενοχικό δίκαιο. Άρα σε όλες τις περιπτώσεις συναλλαγών B2C ε, και B2B υπάρχει κόστος συναλλαγής. Και το διασυνοριακό κόστος ε, οφείλεται στις διαφορές του δικαίου που χώρα σε χώρα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να αποδειχθεί πρώτα απ' όλα ποιο είναι το εύρος αυτού του κόστου συναλλαγής και πώς ορίζονται με αυτόν τον περιοριστικό τρόπο και δεύτερον πώς η πρόταση αυτή αναμένεται να επηρεάσει το κόστος της συναλλαγής, γιατί ο σκοπός είναι να μειωθεί αυτό το κόστος και να αυξηθεί αντίθετα το όφελος από την εναρμόνιση ή την μερική αναρμόνιση. οποιοδήποτε σύστημα ε, προτείνεις, ακόμα και αν είναι προαιρετικό, θα οδηγήσει σε επιπρόσθετο κόστος συναλλαγών, ε, επιπρόσθετο σε σχέση με αυτό που και Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία και μια δυσάτμιση ανάμεσα στο υφιστάμενο κόστος συναλλαγών και αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε με την πιθανή μεταγενέστερη εφαρμογή του νέου προτινόμενου συστήματος. Πώς αντιμετώπισε η Κομισιόν αυτόν τον υπολογισμό. Και εκεί έγινε το, το κύριο πρόβλημα που εμείς έχουμε με αυτή τη μελέτη δικτύπου. Είναι ότι τα δεδομένα που χρησιμοποίησε για να κάνει τον υπολογισμό τα απέσπασε από τρεις πηγές. Πρώτη πηγή είναι η υπηρεσία του βρεβαρόμετρου και οι δύο άλλες πηγές είναι αρκετά περιορισμένες ε, πηγές που είναι ένα πάνελ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα άλλο πάνελ υπητή. E άμα δείτε τα βασικά γράφα λένε ότι αυτά τα, τα πάνελ δεν είναι ε, αντιπροσωπευτικά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλο λοιπόν ένα πρόβλημα. Ευρωβαρόμετρο λοιπόν από τη μία, ε, e και πάνελ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίνουν την ίδια κατεύθυνση ότι οι συνδυσιονικές περιπτώσεις, οι συναλλαγές φέρουν ένα σημαντικό κόστος και επηρεάζεται το κόστος αυτός από τις διαφορές που υπάρχουν στο νοχικό δίκαιο. Και από εκεί και πέρα είναι αδύνατο να υπολογιστεί το εύρος αυτών των διαφορών. Η υπηρεσία του υπερβαρόμετρου ξέρουμε ότι δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες, που σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είναι τα κατάλληλα στοιχεία. Δηλαδή από έτσι αφηρημένες γενικές ερωτήσεις που τίθενται σε μια επιχείρηση τηλεφωνικά, δεν μπορείς να κάνεις μια προβολή τέτοια ώστε να καταλήξεις στα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει μια μελέτη τύπου. Επιστημονικά αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήξαμε και όχι μόνο εμείς, οι μαζικές επικρίσεις εδέχθηκε στη μελλοντική ούτως ή άλλως. Και το δεύτερο ερώτημα που ετέθη, καθώς δεν έμεινε το θέμα εκεί, είναι μπορεί κανείς ε, να τα πάει καλύτερα. Είναι δυνατό να κάνει κανείς μια, έναν καλύτερο υπολογισμό του κόστου ε, των συναλλαγών. Εμεί δεν είμαστε οικονομολόγοι, οπότε απευθυνθήκαμε σε έναν οικονομολόγο, ειδικό και ρωτήσαμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε την μέθοδο της Κομισιόν. Ναι, ήταν η απάντηση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σου δώσει τη συγκεκριμένη φόρμουλα, την εξίσωση με την οποία θα υπολογίσεις το κόστος ε, της συναλλαγής. Οπότε ο επόμενος που θα βρει αυτή την εξίσωση θα πάρει και το επόμενο βραβείο ε, Νόμπελ στα μαθηματικά. Από εκεί και πέρα, πολλά στοιχεία στην πλήρη που δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα υπέρ και τα κατά της πρότασης, αν θέλετε, μας δίνεται για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτή τη μείωση του κόστους των διεθνωτικών συναλλαγών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε πολύ ακριβή και αξιόπιτα ε, στοιχεία. Εκεί θα πρέπει να δουλέψει και ξεκάθαρα η Καμισιόν, ώστε να πει πιο ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και όχι να προσποιείται ότι υπάρχουν δεδομένα και τις επιτρέπουν να κάνει ασφαλείς ε, υπολογισμούς. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μας και με χαρά να μπούμε και σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα, αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ για την ξεκάθαρη παρουσίαση. Δεν κύριο Σάπερμα πρέπει να είχα καλωσορίσει ήταν κάπου κρυμμένος, παλιός ε, φίλος της Επιτροπής μας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές για να δώσουν και τη δική τους πλευρά και τις δικές τους προτάσεις. Η κυρία Γκέπαρτ και μετά ο κύριος Μάιερ θα πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Βανών για την εργασία που ε, προσφέρει πάρα πολλά διδάγματα και είναι σημαντικό που βλέπω οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου να εργάζονται τόσο διεξοδικά και τόσο επιτυχημένα ζητώντας και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και πραγματογνωμοσύνες έξωθεν. Εγώ εξ όσων μας είπατε, συμπεραίνω, ότι η μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις μελέτες αντικτύπου είναι... ήταν καλύτερη από αυτή που έχουμε συνήθως. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό και καλό. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ποια είναι τα ουσιώδη συμπεράσματα και σε ποια βάση εξάγονται τα συμπεράσματα αυτά. Εδώ έρχεται σε ένα από τα δύο σημαντικότερα θέματα της επιχειρηματολογίας της Κομισιόν. Το κόστος των συναλλαγών δηλαδή, που σημειώνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς και το να καταστούν τα προϊόντα για τους καταναλωτές φθηνότερα. Είπατε ότι θα έχουμε και νομπελίστα που θα μας εξηγήσει πώς μπορούμε να υπολογίζουμε το κόστος των συναλλαγών. Άκουσα με ενδιαφέρον στην μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πολλές επιχειρήσεις οι ίδιες δεν γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία κόστους των συναλλαγών τους. Δεν ήταν σε θέση οι ίδιες δηλαδή να δώσουν τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Το δεύτερο μέγα επιχείρημα που ε, το βλέπω πάλι στο έγγραφο της κυρίας Βαρώνη είναι η πτώση των τιμών καταναλωτού αλλά στη σελίδα 107 της μελέτης επιπτώσεων της Κομισιόν διαβάζω της Κομισιόν ξαναλέγω, ε, ξαναλέγω ε, η Διευθυντική Κομισιόν λέει ότι με τον αυξημένο ανταγωνισμό αναμένουμε πτώση των τιμών κατά 0,04 έως 0,07%. Αν αυτό είναι το επιχείρημα για την εισαγωγή ενός απολύτως νέου συστήματος, ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό γίνεται πια γελίο. Θα επανέλθω σε μια άλλη παράθεση, στη σελίδα 26, του πονήματος ε, των υπηρεσιών μας με την αξιολόγηση ε, δύο μόνων επιχειρήσεων και των στοιχείων του Ευρωβαρόμετρου, όπου δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα δεδομένα της, του πεδίου εφαρμογής και αυτό επιτρέπει κάποιες αμφιβολίες για την ορθότητα των δεδομένων της Κομισιόν. Και επίσης δεν λήφθηκε υπόψη και το ότι έχουμε στο μεταξύ την οδηγία των δικαιωμα... του δικαίου των καταναλωτών, έτσι είναι κύριε Σφάπ, που υπάρχει κάποια εναρμόνιση και όπου έχουμε μέσα στην οδηγία καταναλωτών τέτοια εναρμόνιση και όμως επανέρχεται στο σύστημα αυτό που είναι ζήτημα επιλογής μεταξύ κοινοτικού και εθνικού δικαίου και όπου πάλι εκεί το δικαίωμα των, ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν παραλαμβάνονται και αυτό οδηγεί στην ύπαρξη, τριών συστημάτων. Αυτό μπορεί να σημαίνει άραγε ασφάλεια δικαίου, ενώ ακριβώς αυτό είναι το δικό μας καθήκον, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου. Ένα τελευταίο, θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα βέβαια, αλλά βλέπω πόσο έχει προχωρήσει η ώρα. Επίσης λοιπόν ήθελα να πω για την ακρόαση που διεξήχθη χθε για την εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών και να θυμίσω τα όσα είπε ο κ. Πέλκμανς στο πλαίσιο αυτό, ο οποίος είπε ότι το μέγα μειονέκτημα της ενιαίας αγοράς στις υπηρεσίες είναι η ετερογένεια του δικαίου. Αυτή η ετερογένεια του δικαίου, επαναλαμβάνω, και σύστησε ο κ. Πέλκμανς να εργαστούμε περισσότερο προς την κατεύθυνση μιας εναρμόνισης. Αυτά που μας λένε οι δικοί μας, οι εμπειρογνώμονές μας, και ασφαλώς το όργανο δεν είναι ε, κανένα σοσιαλδημοκρατικό όργανο, είναι των επιχειρήσεων. Και όμως μας λέει αυτό τον δρόμο να ακολουθήσουμε. Τώρα, για τον τομέα των ψηφιακών προϊόντων έχουμε την μεγάλη ευκαιρία. Διότι εκεί δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα παρά ελάχιστο, ελάχιστο δίκαιο στις χώρες Εκεί λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί από τα κάτω, από τη βάση δηλαδή, ένα ευρωπαϊκό δίκαιο. Και τέτοιες προτάσεις θα κάνω άλλωστε και εγώ η ίδια. Και Μάιερ. Ναι, σύντομα κι εγώ. Είδα ότι ένευσε καταφατικά ο πρόεδρος μας για την ε, εναρμόνιση. Δεν νομίζω όμως οι Άγγλοι νομικοί να ενθουσιαστούν με την ιδέα να εναρμονίσουμε το common law ε, μέσα στο ε, δίκαιο των συναλλαγών. Ας μείνουμε λοιπόν στο impact assessment. Σήμερα θα δούμε τα υπόλοιπα αργότερα. Ένα πράγμα είναι σαφές. Στην αξιολόγηση αυτής της impact assessment που έχουμε τώρα μπροστά μας, ακούσαμε και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι η ανάλυση της Κομισιόν καταρχήν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, διότι είναι το, το καλύτερο που είναι αυτή τη στιγμή εφικτό. Εάν τώρα πούμε ότι κάποια πράγματα δεν έλαβε υπόψη που υπάρχουν, που είναι επιστημονικά θεμελιωμένα κτλ., τότε αυτά είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να απαιτούμε περισσότερα από την Κομισιόν από όσα επιστημονικά είναι δυνατόν να γίνουν. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι εν πάση περιπτώσει το κόστος των συναλλαγών διαμεθοριακά είναι μεγαλύτερο από ότι μέσα στα πλαίσια μια συγκεκριμένη επικράτεια. Ιδίω όταν προκύπτουν διαφορέ. Γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμά ότι οι καταναλωτέ δεν είναι σε θέση να ξεκινήσουν μια διαδικασία διαμεθοριακή για επίλυση μια διαφορά η οποία θα του κοστίσει εκατοντάδε ευρώ, διότι δεν έχουν δυνατότητα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες δυνατότητες όπως το ευρωπαϊκό small claim, η διαδικασία small claim και ούτω καθεξής. Τώρα, αυτά εξηγούν γιατί οι ε, επιχειρήσεις διστάζουν να δραστηριοποιηθούν διαμεθοριακά. Αυτό είναι όμω ένα λόγο. Η οικονομική συμπεριφορά, ωστόσο, βασίζεται συχνά και σε ψυχολογικού παράγοντε. Ήδη η προσφορά με την έννοια ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα εμπορικό δίκαιο εφόσον υπάρχει και εφόσον το δέχεται και ο, ε, ο, ε, ο άλλος, ήδη αυτό είναι μια επιτυχία. Το ερώτημα περισσότερο είναι όχι τόσο εάν οι καταναλωτές δεν αγοράζουν στο εξωτερικό διότι δεν γνωρίζουν το δίκαιο αυτό που ε, διαθέτουν, αλλά εάν οι πολιτές τους επιτρέπουν, τους προσφέρουν τη δυνατότητα δηλαδή να αγοράζουν σε άλλες χώρες, διότι δεν υπάρχει προσφορά. Επαναλαμβάνω, πηγαίνετε στο διαδίκτυο και προσπαθήστε να αγοράσετε, για παράδειγμα, σε κάποιες από τις νέες χώρες μέλη μας. Θα δείτε ότι καταρχήν αυτό είναι αδύνατο. Εφόσον έχουμε, έχουμε νέα αγορά και ως Επιτροπή Ενιαίας Αγοράς το καθήκον μας είναι αυτό να ανοίξουμε την ενιαία αγορά. Στην ενιαία αγορά λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει προσφορά παντού και να μπορεί να αγοράζει ο καταναλωτής παντού. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή θα έχετε τη δυνατότητα να προβείτε στην αγορά, τότε έρχεται και το δεύτερο μέρος, υπό ποιε προϋποθέσεις, υπό ποιε συνθήκες και όρους μπορείτε να προβείτε στην αγορά ή ενδεχομένως ε, να ε, αμφισβητήσετε ή να ανακαλέσετε και το Αυτό πρέπει λοιπόν να είναι το πρώτο βήμα και ως πρώτο βήμα αυτή η μελέτη αντικτύπου είναι ενδεδειγμένη. Εάν μειώσουν οι επιχειρήσεις το κόστος συναλλαγών, Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς μια επέκταση της ενέας αγοράς. Περί αυτού πρόκειται και για τα επιμέρους ουσιώδη ε, θέματα έχουμε χρόνο ακόμα να τα συζητήσουμε. δεν μίλησα για πλήρη εναρμόνιση, μίλησα για εναρμόνιση απλώς. Εγώ θα επανερχόμουν σε αυτό το σημείο στη συνέχεια, στις καταληκτικές μου παρατηρήσεις ξέχασα να καλωσορίσω και τον κύριο Μπελιγκέρντ από την ε, Επιτροπή, εκπροσωπεί την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Να ακούσουμε πρώτα τα μέλη μα και μετά θα σα δώσω το λόγο. Οι υπόλοιποι σκιώδει, Κύριε Κρόιτσμαν. Εναρμόνιση, καλή είναι η εναρμόνιση, αλλά όπως γνωρίζετε τα δαιμόνια κρύβονται στι λεπτομέρειε. σε ποιο επίπεδο θα κινηθεί η εναρμόνιση, στο ύψιστο επίπεδο, στο χαμηλότερο, ιδίω για θέματα καταναλωτών, η Γερμανία έχει σχετικά υψηλό επίπεδο. Αν ε, μειώσει το επίπεδο αυτό, τότε θα αρχίσουν όλοι να φωνάζουν. Ο κύριος Μάιερ είπε προηγουμένως για νομολογία ε, και το ε, common law απέναντι στο, σε αντιπαράθεση δηλαδή με το ρωμαϊκό δίκαιο. Το κοινό εμπορικό δίκαιο, εάν είναι εθελοντικό, θα έχει την ευκαιρία να ε, κυριαρχήσει συν το χρόνο και να οδηγήσει επομένως σε μεγαλύτερη αναρμόνιση. Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, περισσότεροι συμμετέχοντες, άρα ευνοϊκότερο για τους καταναλωτές, χαμηλότερα κόστη συναλλαγών για τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά όμως ως λιδία λίθο έχουν την εμπιστοσύνη. Αν θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή τα πράγματα αυτά, οι δυνατότητες αυτές, ή αν θα πούν, α, καλύτερα για να είμαι σίγουρος να πάω στον έμπορο επιτόπ. Και τώρα για την μελέτη αντικτύπου που πιστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δούλεψε καλά και καθαρά. Αυτό είναι σημαντικό. Δείχνει και, τις, και τα δύναμα σημεία. Δεν μπορούν βέβαια όλα να ποσοτικοποιούνται εάν όντως το πλεονέκτημα θα είναι της τάξης του 0,045% κυρία Κέπχαρτ, έχετε δίκιο. Ωστόσο, αν υπάρξουν και άλλα ωφελήματα, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, πολλές επιφυλάξεις στη Γερμανία από πολλές πλευρές, αλλά στο κάτω της γραφής κανένας δεν υποχρεούται να το εφαρμόσει. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να γίνει η προσπάθεια. Θα μπορέσει, πιστεύω, να ενισχύσει την ενιαγορά, μπορεί να αποβεί προς όφελος του καταναλωτού και αν είναι μετρήσιμο το όφελος, τότε πράγματι αξίζει τον κόπο να γίνει μια προσπάθεια για ένα κοινό ε, εμπορικό δίκαιο. Βέβαια, μπορεί να λυθεί το θέμα με ένα νομοθέτημα μερικών σελίδων. Θα είναι μικρότερο από το γερμανικό αστικό κώδικα. Αλλά παρόλα αυτά είναι μέγα έργο. Είναι λοιπόν διατεθειμένος κανείς, και Επχαρτ, ο ενδιαφερόμενος δηλαδή, να εγκαταλείψει τα όσα γνωρίζει και να πάει να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο του είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο. Έχω κάποιες αμφιβολίες, διότι οι καταναλωτές συνήθως στρέφονται σε αυτά τα οποία τους είναι ήδη γνωστά και αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο να καλέσω από του συναδέλφου να είναι εξαιρετικά σύντομοι, γιατί ε, βρισκόμαστε στην αρχή της συζήτηση, όχι στο τέλος. Ε, Πρώτα, ευχαριστώ ιδίω τι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και απευθύνω έκκληση στην Κομισιόν να συναγάγει τα συμπεράσματά της, ώστε στο μέλλον να είναι πιο ρεαλιστική, γιατί συχνά μας υποβάλλει μελέτες αντικτύπου που υπόσχονται τα πάντα εγώ στις ε, σπουδές μου έκανα και μαθήματα συγκριτικών στατιστικών και βλέποντας κάτι τέτοια πράγματα πραγματικά μου αναστατώνεται το στομάχι, πώς να σου το πω. Αυτή λοιπόν είναι η κρίση μου, κάπως μεγαλύτερη σοβαρότητα με αυτές τις impact studies και με τις υποτιθέμενες εξοικονομήσεις κόστους. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση, μόλις αρχίσαμε. Κύριε Κρότσμαν, εξακολουθούμε να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το αν θα αποφέρει τίποτα αυτό το εθελοντικό καθεστώς. Και θα θέλαμε η Κομισιόν να περιμένει να δει τι θα αποδώσει η ε, Οδηγία Προστασίας των Καταναλωτών και να κάνει τα, επόμενα βήματα. Κύριε Παναγιά, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για την Επιτροπή, από την πλευρά της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε αυτό το προνόμιο να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας και θα πω μόνο το εξή Στην Επιτροπή Γιούρη, ο συνάδελφος λένε και εγώ, υποβάλαμε χθες το σχέδιο έκθεσης μας για το θέμα αυτό. Αυτό το σχέδιο έκθεσης βασίζεται και στη μελέτη αντικτύπου και φυσικά στην πρόταση της Κομισιόν. Προτείναμε ένα ψηλό αριθμό τροπολογιών, οπότε αν εγκριθεί η έκθεσή μας, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει τροποποιηθεί ριζοσπαστικά. Είμαστε πεπισμένοι ότι είναι γεμάτο λατώματα το κείμενο της Κομισιόν. Επιλέξαμε όμως ένα δρόμο βασιζόμενοι σε προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας. Δηλαδή, να επιλέξουμε το optional instrument, ότι είναι ένα προαιρετικό εργαλείο αυτή η οδηγία. Η εναρμόνιση επελέγει βάσει του οδηγού των καταναλωτών, αλλά αποδεικνύεται ανεπαρκής. Είναι δίνει τα ελάχιστα, αλλά είναι ανεπαρκής. Σήμερα η προστασία του καταναλωτή διασυνοριακά είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί? Γιατί περιορίζεται μόνο σε αυτό, χωρίς να δημιουργεί μία δυνατότητα ε, συνθήκων ώστε να έχει πρόσβαση σε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς του καταναλωτάς και άρα να εγγυηθεί την ουσία του δικαίου. Χαμηλές τιμές, υψηλή ποιότητα, μεγαλύτερη προσφορά. Αν λοιπόν δεν δείξουμε αποφασιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, τελικά τι κάνουμε. θα προωθήσουμε κάτι που δεν έχει πόδια να σταθεί. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει άρδιν το κείμενο της Κομισιόν. Και γι' αυτό θέλουμε μια επαφή ανάμεσα στις δύο Επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να δουλεύουμε παράλληλα, αλλά μαζί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και εργασίες της δικής της Επιτροπής. Χρειαζόμαστε λοιπόν τις επαφές μαζί σας, ώστε οι αλλαγές που θα γίνουν στην πρώτη Κομισιόν να μπορούν να εγγυηθούν ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την πρόσταση του καταναλωτή και για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε εδώ. Συγγνώμη που δεν σας είχαμε δώσει το λόγο προηγουμένως για την αξιολόγηση δικτύπου. Θα περιμένουμε τα... την έκθεση των δικών μας εισηγητών. Α, να προσθέσω μόνο μια λέξη. Και κάτι ακόμη. Η πιο σημαντική αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι ότι περιορίσαμε το πεδίο εφαρμογή μόνο στις ε, επιγραμμικές συμβάσεις και τις τηλεσυμβάσεις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και με πέντε χρόνια α, επαλήθευσης τουλάχιστον θα ε, κινητοποιηθεί, θα δημιουργηθεί και θα κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός για να δούμε πού μπορούμε να πάμε καλύτερα. Σημαντική είναι αυτή η αλλαγή. Και ειλικρινά μόνο και μόνο για αυτή τη σημαντική αλλαγή απαιτείται περαιτέρω ανάλυση, γιατί αλλάζει τη βάση αυτού του οικοδομήματος. Γιατί ο υπολογισμός του συναλλαγματικού κόστος, το κόστος των συναλλαγών μάλλον, ε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Το δικό μου πρόβλημα, ε, το οποίο εντοπίζω, είναι ότι σε αντίθεση με τις κατευθυντήρες γραμμές ε, της Επιτροπής, το πρόβλημα αυτό δεν είναι συμπεριλαμβάνει το σενάριο που θα περιγράφει πώς ακριβώς θα, καθοριστούν οι βασικές γραμμές χωρίς ενέργειες. Και υπάρχει, απορρίπτεται μάλλον η ε, λύση της αδράνειας, το να μην κάνουμε τίποτα δηλαδή. Είναι ενδιαφέρουσε οι ιδέες αυτές, όμως το κόστος ε, ίσως να είναι μεγαλύτερο από το όφελος. Γι' αυτό θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Δεύτερον, εξαρτάται το πόσοι θα επιλέξουν ε, αυτό το δρόμο ευθύ εξ αρχή. Δεν υπάρχει όμω καμία ένδειξη για το πώ ακριβώ θα κάνουν αυτή την επιλογή και για να δούμε και τι εξοικονομήσει ε, δαπανών. Και τρίτον, μεθοδολογικό σφάλμα δεν είναι σαφέ, δεν υπάρχει σαφή ένδειξη για τη σχετική σημασία της έλλειψης εναρμόνισης ε, στους συμβατικούς όρους σε σχέση με άλλα θέματα που αντιμετωπίζει κάποιο κατά τη ε, διασυνοριακή συναλλαγή. Και τα δεδομένα ε, ε, δεν είναι καταλεκτικά. Δεν μας βοηθούν δηλαδή να συναγάγουμε συμπεράσματα. Βεβαίως έχουν γίνει βήματα στο παρελθόν, όμως έχει περάσει ο καιρός. Σίγουρα λοιπόν θα γίνει στη δουλειά του συζητητέ. Όμω καλά κάνει η κυρία Γκέπχαρτ και αναφέρει τα όσα λέει. Ότι δηλαδή η δυνατότητα ύπαρξης εναρμονισμένων νόμων, όχι απαραίτητα με την πλήρη εναρμόνιση, αλλά θα αποτελούσε ένα σημαντικό όφελος ε, για την οικονομική δραστηριότητα. Έχουν τεθεί επιτάπητος οι εναρμονισμένοι νόμοι για τα δικαιώματα καταναλωτών, ε, έχουν εφαρμοστεί και με θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ιδέα και ενό ε, τυποποιημένου, μιας τυποποιημένης σύμβασης, ενός συμβολέου που θα μπορούσε να ε, χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Ίσως θα πρέπει να την εξετάσουμε. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει εναλλακτική λύση ε, στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο ε, διαδικτυακών συναλλαγών. Αυτέ είναι οι δικές μου παρατηρήσεις. Δεν είμαι ούτε καν ω εισηγητή, δεν τις κάνω, ούτε καν ω σκιώδη, αλλά ως ε, πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους για τη συμμετοχή σας. Ε, περιμένουμε ε, την έκθεσή σας και θα επανέλθουμε στις 3 ε, το απόγευμα. Ευχαριστώ.